So good morning, <laughs> one more colleague. So we can uh, start and of course we have a meeting with the national. Um, Προβλέπετε να κάνουμε μια συνάντηση με τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχουμε όμως διάφορα υπόλοιπα από την ε, προηγούμενη συνεδρίασή μας και δεν είναι πολλοί συνάδελφοι παρόντες αλλά μπορούμε να εγκρίνουμε ίσως την ημερήσια διάταξη και θέλω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Ως πρόεδρος συνάντησα <clears throat> τον ε, εισηγητή του των Ηνωμένων Εθνών για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, τη συμφιλίωση και τη μη επανάληψη των διαμαχών. Αυτό είναι μια, ένα αξίωμα το οποίο δημιουργήθηκε πρόσφατα και προσπαθεί ο εισηγητής αυτός των ΗΠΑ να εξασφαλίσει όλα τα στοιχεία της μεταβατικής δικαιοσύνης να ληφθούν υπόψη. και να θέλει να εξασφαλίσει την ε, λογοδοσία και την ε, συμφιλίωση, να υπάρξει ανεξάρτητη εποπτεία του συστήματος ασφαλείας, να επανέλθει η εμπιστοσύνη στο, στους κατοικούς μηχανισμούς και να προωθηθεί το κράτος δικαίου βάσει των διεθνών προτύπων. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Είπε ότι σε όλους αυτούς τους τομείς η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ως ένας παγκόσμιος παίκτη για τα θέματα αυτά, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε ακόμα δυσκολίες να είμαστε συνεκτικοί στις ε, ε, πρωτοβουλίες αυτές. Ίσως λοιπόν κάποιος βουλευτής θα βρει την ευκαιρία να κάνει μια έκθεση πρωτοβουλίας και να δει σε ποια από αυτά τα εργαλεία πρέπει να κάνουμε προσπάθειες για να προωθήσουμε περισσότερο την δικαιοσύνη, την αλήθεια και τη συμφιλίωση. Επίσης, ο... Ο βραβευμένος με το βραβείο 2008 είναι σε κατοίκον κράτηση και πρέπει η Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης να δώσει συνέχεια με μια διαμαρτυρία για το θέμα αυτό. Πρέπει να ανακοινώσω επίσης ότι θα έχουμε η Aung San Suu θα είναι μαζί μας τον Οκτώβριο όπου θα λάβει επιτέλους το βραβείο Σαχάροφ. 21 Οκτωβρίου θα είναι μαζί μας. Έχουμε μια κοινή συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την 3η 22 Οκτωβρίου θα έχουμε μια συνάντηση μόνο μαζί της στην Ολομέλεια. Για τον Μπαχρέιν. Ο κ. Χαλίλ Αλμασούκ, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Μεγάλου ε, κόμματος αντιπολίτευσης Αλρεφάκ ανακρίθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου από τον ανακριτή και παραμένει για 30 μέρες στη φυλακή κατά τη διάρκεια των ερευνών. Τον ανακρίναν σε σχέση με τα γεγονότα της 6 Σεπτεμβρίου όταν οργάνωσαν ένα συλλαλητήριο δυνάμεις της αντιπολίτευσης με παρουσία 6.000 ατόμων. Ο κ. Χαλίλ Αλμασούκ είχε λάβει το λόγο σε αυτή τη συγκέντρωση. Είμαστε και <clears throat> πάλι σε επαφή με την, Ευρω... με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τα θέματα αυτά. Επίσης, μία από, τις, ε, ε, μία από τα μέλη της, ε, του Pussy Riot στην, στη Ρωσία έχει ξεκινήσει μια απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθεί για τις συνθήκες σκλαβιάς στη φυλακή όπου εκτείνει μια ποινή δύο ετών. Και επίσης, να συνεχίσω από την προηγούμενη από την προηγούμενη συνεδρία μιλήσαμε για την ε, καταναγκαστική εργασία στο Καζακστάν σε σχέση με τη συλλογή ε, Βάμβακος και είχαμε και τη μαρτυρία ενός ατόμου από το Καζακστάν ο οποίος έμεινε κρατούμενος στο Ουργέν στην ε, πόλη του και έχει απαγορευτεί η επαφή του με οποιονδήποτε. Έχω συντάξει μια επιστολή λοιπόν <clears throat> προς τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την Κεντρική Ασία για να δώσει συνέχεια στα θέματα αυτά. Αυτά λοιπόν για τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Και τώρα έχουμε την έκθεση από την επίσκεψή μας στην Αφρικανική Ένωση και την Αιθιοπία. Δυστυχώς δεν ήταν κανένας εδώ από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και γι' αυτό χρειάζεται να επανέλθουμε στη σημερινή συνεδρίαση. Έδωσα μία πλήρη έκθεση για τα θέματα αυτά. Αλλά ο κύριος Βίσεπ έθεσε ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με την απεργία πείνας του δημοσιογράφου Αλέμου και θέλουμε να ξέρουμε από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αντισαμπέμπα ποια είναι η κατάσταση του δημοσιογράφου αυτού και τι συνέχεια έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αυτά. Ξέρετε ότι εμείς είχαμε σκοπό να επισκεφθούμε τη φυλακή Καλίτη στην ε, Αντισαμπέμπα και να επισκεφθούμε και ορισμένου από τους αρθογράφου στο διαδίκτυο bloggers οι οποίοι κρατούνται εκεί. Μας είπε ο Διευθυντής φυλακή ότι δεν έχει χρόνο να μας δείξει τη φυλακή ή να μας επιτρέψει να συναντηθούμε με, τα, με τους κρατούμενους αυτούς. Μία από τις προτάσεις που είχαμε κάνει τότε στον Διευθυντή των Φυλακών είναι αν υπήρχε χρόνο στις ε, επόμενες ημέρες να μπορέσει η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επισκεφθεί τη φυλακή. Αυτό έγινε με την ε, κατανόηση ότι ο επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας που θα ήταν παρόν και αυτός, γιατί και αυτός εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι μας εκδίωξαν από τη φυλακή. Ο κ. Βησέ επίσης θέλει να ξέρει περισσότερο για το πρόγραμμα της εγκατάστασης σε χωριά σε ορισμένες πολύ φτωχές περιοχές. Πρόκειται για εγκατάσταση, επανεγκατάσταση νομαδικών πληθυσμών σε πάρα πολύ φτωχές περιοχές και φαίνεται ότι όταν ήμασταν εκεί είπαν ορισμένοι εκπρόσωποι αυτών των νομαδικών κοινοτήτων ότι κανείς δεν έχει ζητήσει τη γνώμη τους αν θέλουν να εγκατασταθούν με αυτόν τον τρόπο σε χωριά ή κάτω από ποιες συνθήκες θα θέλανε να εγκατασταθούν. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε πώς έχει προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα. Κάποιες από τις διεθνείς ΜΚΟ μας δίνουν ε, αναφορές ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των νομαδικών κοινοτήτων βοσκών έχουν ε, κατά πάσα πιθανότητα παραβιαστεί. Εάν θέλετε λοιπόν να κάνετε κάποια σχόλια για αυτές τις εκθέσεις, γιατί μας είπαν τότε οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων, αλλά και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι, <clears throat> ότι υπάρχουν αυτές οι εκθέσεις και ανακοινώθηκε ότι θα υπήρχαν και νέες εκθέσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα θέματα αυτά. Αυτά λοιπόν. Η κυρία Γκυγέμ τώρα που είναι η αρμόδια για τα θέματα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Hello everyone. Um, apologies for last... Συγγνώμη για την περασμένη εβδομάδα. Είχα να αντιμετωπίσω μια πιούσα κατάσταση και δεν μπορούσα να έρθω. Χίλια συγγνώμη. Καλημέρα σε όλους. Το καλό είναι βέβαια ότι είχα τη δυνατότητα να έχω απαντήσεις από την αντιπροσωπεία επιτόπου για τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ λοιπόν που μου τα μεταφέρατε. Όπως γνωρίζετε, κάναμε μία συνάντηση τον Ιανουάριο προπαρασκευαστική για την ε, ε, δική σας επιτροπή, για την επίσκεψη της δικής σας επιτροπής. Παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία. Όσον αφορά την κατάσταση των, του Ηματαλέμου, του δημοσιογράφου, προσπαθούμε να τη χειριστούμε, να την παρακολουθήσουμε όσο το δυνατόν πιο ε, στενά ή ε, δημοσιογράφος, συγγνώμη, ε, η οικογένειά της μας είπε ότι δεν, είναι, δεν κάνει πλέον απεργία πείνας, τη σταμάτησε. Ζητήσαμε από την αιθιοπική κυβέρνηση να δώσει τη δυνατότητα επισκέψεων στην οικογένειά της. Καταλαβαίνετε ότι είναι δικαίωμα αναντήρητο για όλους τους ε, κρατουμένους. Όσον αφορά τώρα την επίσκεψη στη φυλακή, λάβαμε επιβεβαίωση ότι οποιαδήποτε επίσκεψη σε σχέση με την αναθεώρηση των συνδικών κράτη φυλακές ε, είναι δυνατή. Η αντιπροσωπεία είχε τη δυνατότητα να συναντήσει τη διεύθυνση των φυλακών. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ποια ημερομηνία ε, ε, θα γίνει αυτό και μετά θα γίνει η επίσκεψη και των φυλακών. Η επίσκεψη των Ευρωβουλευτών ακυρώθηκε επειδή θεώρησε η αιθιοπική κυβέρνηση ότι άλλαξε ο στόχος της από την αναθεώρηση των συνθηκών στις φυλακές ε, στην επίσκεψη της συγκεκριμένης δημοσιογράφου. Και όπως γνωρίζετε η κυβέρνηση της Αιθιοπίας ε, έχει τη θέση ότι δεν είναι πολιτική δεν έχει πολιτικούς ε, κρατούμενους και γι' αυτό ακριβώς δεν θέλει να ξεχωρίσει κανέναν ε, κρατούμενο. Όταν λοιπόν ζητήθηκε η επίσκεψη της συγκεκριμένη ε, κρατούμενης, αποφάσισαν να κυρώσουν την επίσκεψη. Βεβαίως κρίμα, όπως είπατε κι εσείς. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση ε, μας ε, επιβεβαίωσε ότι μπορεί να γίνει επίσκεψη ανα πάσα στιγμή για την αναθεώρηση των συνθηκών κράτησης φυλακές ε, και για την ενίσχυση ε, της προσπάθειας κυβέρνησης ε, για τη βελτίωση των συνθηκών αυτών. Επίσης λάβαμε πληροφορίες ότι από την αρχή το 2013 ε, είχαμε άμεση πρόσβαση ε, σε όλους τους κρατουμένους ε, και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο και επομένως τουλάχιστον η συνεργασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο συγκεκριμένο θέμα έχει βελτιωθεί από τις αρχές του έτους. Σε γενικότερες γραμμές τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με την εφαρμογή, ενδιαφέρεται με την εφαρμογή της αντιτρομοκρατικής ε, ε, πολιτικής με την οποία ασχολήθηκε η δημοσιογράφος που κρατείται, κάτι το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 ε, του πολιτικού μας διαλόγου και συζητήθηκε το Δεκέμβριο του 2012 με τον Πρωθυπουργό. Όσον αφορά τώρα την εγκατάσταση στη χωριά και το σχετικό πρόγραμμα, μπορούμε να ε, σας ενημερώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δεν χρηματοδοτούν το πρόγραμμα αυτό ε, της αιθιοπία. Ε, από το 2010 όμως, δωρητές της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, ε, μέλος ε, των διεθνών δωρητών για την Αιθιοπία, έχουν ένα διάλογο με την κυβέρνηση για θέματα μεταξύ των οποίων τη βελτίωση της εφαρμογής του προγράμματος αυτού, καλύτερες κατευθυντήριες γραμμές, όπως επίσης και μηχανισμούς αποκατάστασης. Και από το 2011 οι δωρητές συμμετείχαν σε τουλάχιστον 10 αποστολές ε, δωρεών ε, ειδικότερα για το πρόγραμμα εγκατάστασης ε, σε χωριά και άλλα σχετικά προγράμματα. Θα υπάρξουν νέες εξελίξεις και αυτή τη χρονιά. Δεν έχουμε καταφέρει να στοιχειοθετήσουμε ισχυρισμούς για κατάφορες παραδιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν, υπήρχε κάποια παρεμπόδιση με την κατάσταση ε, πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ε, πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Ε, εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τις, την κατάσταση μέσω του άρθρου 8. Ο Υπουργό Ανάπτυξη επίση είναι σε συνεργασία μαζί μα ε, για τέτοιου είδου προγράμματα. Εμεί είμαστε ε, διατεθειμένοι να συνεχίσουμε το διάλογο με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία των πολιτών. Η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα εξακολουθήσει να αποτελεί ένα τμήμα σημαντικό τη αναπτυξιακή μα ε, συνεργασία με την Αιθιοπία. Ευχαριστώ. Thank you. Are there further... ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις? Ναι. Όχι. Να σας ενημερώσω ίσως ότι αυτό το συζητήσαμε με την Αφρικανική Ένωση Ιδιαίτερα με την ε, Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών ε, για την Οικονομική Ανάπτυξη στην Αφρικανική Ανική Ένωση και συστάθηκε ένα πάνελ υψηλό βαθμό με τη συμμετοχή του πρόεδρου, πρώην Πρόεδρου Μπέκη σε ό,τι αφορά αυτές τις ε, παράνομες ροές χρημάτων έξω από την Αφρική. Και ε, συζητήθηκαν οι πολιτικές και εκδηλώθηκε επιθυμία να ενημερωθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα γίνει στον ΕΟΣΑ η πρώτη ε, ενημέρωση στο Παρίσι. Καταρχάς θεωρήσαμε ότι ενδεχομένως να μπορούσαν να έρθουν και σε εμάς, αλλά είναι πράσινη εβδομάδα. Η Επιτροπή ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ έχουν σχετικά σώματα, μιας και ασχολούνται με θέματα χρηματοδότησης εξωτερικών υποθέσεων και με χρηματοδοτικά. Θα διοργανώσουν μια ακρόαση, θα συμμετάσχει ενδεχομένω και ο Μπέκη. Καλό θα είναι λοιπόν να συμμετέχει και κάποιο από την υπηρεσία εξωτερική δράση που παρακολουθεί το θέμα. Και αυτό παρακαλώ να το μεταβιβάσετε στην υπηρεσία σα. Έχουμε μία γραπτή έκθεση σε σχέση με την αποστολή αυτή. Λάβαμε και κάποια σχόλια. Τα ενσωματώσαμε στην έκθεση. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε πλέον να την ε, μοιράσουμε στα μέλη. Ωραία. Ε, μέχρι τις 10 έχουμε πολύ ώρα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και στις 10 ξεκινάμε την συνάντηση, τη συνεδρίαση. Δεν ξέρω. Γιατί δεν μπόρεσε κανείς να παρευρεθεί. την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί καλό θα ήταν να τα κάνουμε πάντα όλα αυτά μαζί. Ήταν και εκπρόσωπος της πρεσβείας της Αιθιοπίας τότε μαζί μας. Να κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα και ξαναξεκινάμε στις 10 πάλι τη συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Colleagues, I would like to welcome Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας καλωσορίσω όλους. Βλέπουμε ότι υπάρχει συνεργασία Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βλέπουμε πολλά άτομα τα οποία μας είναι γνωστά και άτομα τα οποία μοιάζουν σαν δίδυμοι αδελφοί επίσης, αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Έχει γίνει τακτική, ε, έχουν γίνει τακτικές αυτές οι εκδηλώσεις οι κοινές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εθνικού Κοινοβουλίου και θεωρούμε όλοι ότι είναι αυτό πολύ χρήσιμο. Στην τελευταία συνάντηση του Βίλνιους αντιμετωπίσαμε πολύ δύσκολα θέματα, αλλά μπορέσαμε να βρούμε κοινέ θέσει με μεγάλη ευκολία. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Ξέρετε ότι η εξωτερική πολιτική παραμένει σχεδόν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Συμβουλίου και της Κομισιόν με μικρή συμμετοχή του Κοινοβουλίου, αλλά μετά από τη Συνδίκη Λισαβόνας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντικές νομοθετικές αρμοδιότητες και ένα σημαντικό ρόλο στο δημοκρατικό έλεγχο. Και αυτό καταδεικνύεται σε, από το έργο μας για τα προγράμματα οικονομικής υποστήριξης, από την, ε, από την σύναψη κοινωνικού χαρακτήρα συμφωνιών με τους εταίρους μας. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν το σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε πλαίσια όλων συζητήσεων είναι τα ζητήματα δημοκρατίας, και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως λέω και στο σχέδιο εκθεσής μας, αυτό μας ενδιαφέρει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων μας και φυσικά της υποστήριξης των αξιών μας. Αυτό είναι ένα κλασικό ερώτημα και δίλημα πολλές φορές στην εξωτερική πολιτική, πώς μπορεί κανείς να μπορέσει να εξισορροπήσει τα στρατηγικά συμφέροντα με την διασφάλιση των αξιών. Πολλές φορές έχουμε την εντύπωση ότι μιλάμε περισσότερο για δημοκρατία και ξεχνάμε τα συμφέροντά μας. Άλλες φορές γίνεται το αντίθετο. Και είτε έχουμε real είτε το αντίθετο. Αλλά αυτά είναι, αυτό είναι από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν σήμερα. Και αυτό είναι και ένα από τα θέματα που ε, απασχολεί την Επιτροπή, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με επικεφαλή στην κυρία Λόχμπιλντερ. Ένα από τα κύρια θέματα που μας έχουν απασχολήσει στην έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία είναι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται αυτές τις πολιτικές. Με την ε, έγκριση του πακέτου για την ε, δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκομίσει για πρώτη φορά ένα συνεκτικό πλαίσιο για τα θέματα αυτά. Ο παλιός μας συνάδελφος Σταύρος Λαυρινίδης είναι ο πρώτος <clears throat> εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό καταδεικνύει και τη θέληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ένας παγκόσμιος παίκτης στα ζητήματα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ένας χώρος όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα σημαντικό ρόλο προωθώντας τις αξίες αυτές που την διέπουν από την αρχική της ίδρυση. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η σχέση μας με τους ε, στατηγικούς μας εταίρους η ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής σε εμπορικό επίπεδο συμπεριλαμβάνει πάντα τα θέματα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό είναι πάντα μια κεφαλαιώδης πτυχή. Πολλές φορές αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα και απαιτούμενα για μια εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσπαθήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερα να δώσουμε ένα στρατηγικό πλαίσιο στα θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και λέει αυτό το πλαίσιο ότι ακόμα και έξω από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κοινή ευθύνη των κρατών μελών και τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το στρατηγικό αυτό πλαίσιο θέτει στο επίκεντρο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλες τις χώρες και αυτό συμπεριλαμβάνει και τους στρατηγικού εταίρους τη. Όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στις αρμοδιότητες που τους δίνει η συνθήκη τη Λισαβόνας θα πρέπει να διαδραματίσουν το ρόλο τους για να εξασφαλίσουν την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά μέσα στα πλαίσια μιας κοινή ευθύνη για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του κοινού αυτού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υλοποίησή του σε ένα σχέδιο δράσης και η πρόθεση συγκεκριμένων ενεργειών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα έχουμε μια καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Μπάρμπαρα Λοχμπίλντερ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ να σας καλωσορίσω όλους. Είναι ήδη μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι είναι εδώ μέλη 19 εθνικών κοινοβουλίων και ελπίζουμε να έχουμε μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων. Κάποια από τα κοινοβούλια, η Αυστρία ε, είναι σε προεκλογική περίοδο, η Γερμανία μόλις ε, είχε εκλογές, ε, οπότε θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι οι εκπρόσωποι των κοινοβουλίων εδώ για να μεταφέρουν το μήνυμα που θα ακούσουν ε, ε, πίσω στη χώρα τους. Η αντιπροσωπεία της Λετωνίας δεν έχει έρθει ακόμη γιατί λόγω μίχλης ε, δεν έχει μπορέσει να φτάσει ακόμα. Ελπίζουμε όμως ότι θα έρθουν. Όπως ε, είπε και ο Έλμαρ Μπρόκ, έχουμε ένα στρατηγικό πλαίσιο και ένα σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μας βοηθά πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθήσουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν αναρωτιόμαστε ποιο πρέπει να είναι το θέμα της ανταλλαγής απόψεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια φέτος, θεωρήσαμε ότι ήταν καλύτερα να εστιαστούμε στο πλαίσιο αυτό, ε, και στο τραγικό πλαίσιο για, την, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί όλοι πρέπει να συνεργαστούμε για να το εφαρμόσουμε, που σημαίνει ότι όλα τα κρατημέλη πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η στρατηγική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σωστά μόνο αν ε, ασχοληθούν ε, και τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν χρειάζεται λοιπόν ε, να σας ε, επαναλάβω ότι πρέπει να επενθυμίζουν τα Εθνικά Κοινοβούλια στις κυβερνήσεις ότι πρέπει να επιμένουν στην εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Ε, ο διορισμός του κυρίου Λαμπρινίδη, όπως επίσης και η εφαρμογή των ε, κειμένων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι πολύ σημαντικά ε, για, την εξωτερική, για τις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έτσι στην εκπροσώπησή μας σε διεθνή φόρα τονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά και έχει πολύ πιο ενεργό ρόλο ε, στην προαγωγή ε, των θεμάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, στο σχέδιο δράσης και η στρατηγική ορίζουν σαφέστατα τις ευθύνες είναι λοιπόν πολύ καλό για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δούμε πού έχει φτάσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ε, κατά πόσο ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα ή ε, έχουν καθυστερήσει. Είναι λοιπόν ένα καλό μέσο για μας στο Κοινοβούλιο, ε, ώστε να παρακολουθούμε τι κάνουν. 36 δράσεις, σε, 36 δράσεις ε, και 97 ε, θέματα, εκ των οποίων τα 56 ε, αφορούν και τα εθνικά κοινοβούλια ως προς την εφαρμογή τους, κάτι που μας δίνει μία ακόμη δυνατότητα να δούμε τι ακριβώς έχει δεσμευθεί η κάθε κυβέρνηση να κάνει. Μπορούμε να ρωτήσουμε έτσι και τα εθνικά κοινοβούλια πόσο πολύ έχουν προχωρήσει. Στο Κοινοβούλιο έχουμε μία ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Και ως προς τη δομή της της αυτής της έκθεσης ε, ασχολούμαστε και με την εφαρμογή του, της στρατηγικής. Ο κύριος Κούκαν είναι ο εισηγητής μας και θα, μας, ε, θα παρουσιάσει μέχρι το Δεκέμβριο ένα, ένα σχέδιο δράσης από πλευράς Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε να ακούσουμε συστάσεις και από τη δική σας πλευρά, από την πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων, για να μπορέσουμε να τις συμπεριλάβουμε στην ε, ετήσια μας έκθεση. Έχουμε χωρίσει τη σημερινή μας ε, συνεδρίαση σε δύο συνεδρίες. Πρώτον, ε, στρατηγικό, στρατηγική και ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα ακούσουμε και την τοποθέτηση του Σταύρου Λαμπρινίδη και το απόγευμα θα ασχοληθούμε με την εσωτερική και εξωτερική συνοχή της πολιτικής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι μαζί μας ε, ο κύριος Τόιρμαν που είναι ο πρόεδρος του, ε, της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα είναι και εμπειρογνώμονες ε, από την ε, ΕΕΔ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Κοινωνία των Πολιτών, από οργανισμούς προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκπροσώπους από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Θα έχουμε δηλαδή πάρα πολλές ε, απόψεις, οι οποίες θα ακούσουμε για να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής και ελπίζουμε ότι όλοι σας ε, θα συμμετέχετε ενεργά στη συζήτηση. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λαμπρινίδη για να μας ενημερώσει ε, για τη δουλειά του, όπως επίσης και για τη στρατηγική. Σας ευχαριστώ Μπάρμπαρα και θα ήθελα πραγματικά να σας συγχαρώ για την πάρα πολύ σημαντική αυτή συνεδρίαση. Γιατί όντως, όπως είπατε και οι δύο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν θέλουμε να επιβληθούν πραγματικά σε όλο τον κόσμο, χρειάζονται εταιρική σχέση και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα. Αυτό αποτελεί μία πρόκληση, αλλά και σε ό,τι αφορά την εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών τη κοινοβούλια κράτη-μέλη, ιδιαίτερα πριν τη Λισαβόνα, αγνοούσαν ότι είχαν ληφθεί νόμοι, ότι είχαν πράσει νόμοι σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα όμως ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων ε, ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων έχει αναβαθμιστεί και γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σημαντικό. Τότε, πριν από ένα χρόνο, 27 κράτη-μέλη ε, ενέκριναν ένα στρατηγικό σχέδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάρα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Θεωρώ ότι το έχετε διαβάσει, αν όχι να το διαβάσετε. Αποτελεί ένα παράδειγμα για το πώς 27 κρατη μπορούν να σπάσουν, αν θέλετε, τα ταμπούν και να φτάσουν στον ε, υψηλότερο κοινό παρανομαστή σε ό,τι αφορά μία πολιτική και όχι τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή όπως συχνά θεωρούμε δεδομένο. Επίσης, ενεκρίθηκε ένα σχέδιο δράσεως με 97 συγκεκριμένες δράσεις και οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν και από τα κράτη-μέλη προκειμένου το σχέδιο δράσης να καταστεί αποτελεσματικό. Άρα αναγνώρισαν ότι είναι δύσκολο να υπάρχει ένα φιλόδοξο έγγραφο το οποίο να μην σημαίνει τίποτα γιατί πρέπει να δεσμευόμαστε όχι στο χαμηλότερο δυνατό τεχνικό επίπεδο και πολιτικό επίπεδο. Και τέλος, ε, ορίστηκε ένας ε, υπότος αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ήταν μεγάλη μου τιμή ότι ανέλαβα τα καθήκοντα αυτά. Νομίζω ότι, μια και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, αντί να σας δώσω και να κάνω γενικές παρατηρήσεις για τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πιο σημαντικό θα ήταν να τονίσω τρεις βασικές προκλήσεις τις οποίες θεωρώ ότι αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Αναμφίβολα, είναι σημαντική η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να σκεφτούμε τις συγκρούσεις σήμερα στον κόσμο. Ε, για παράδειγμα, σήμερα ε, στα πλαίσια του ΟΑΣΕ ε, εξετάσαμε κάποια τέτοια θέματα συγκρούσεων, η ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μία οργάνωση. Γιατί, γιατί κοιτάζοντα οποιαδήποτε σύγκρουση σήμερα έναν τον κόσμο, διαπιστώνουμε ότι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνήθω αποτελεί την πηγή, τη ρίζα των προβλημάτων και των συγκρούσεων. Ή η επίλυση ε, παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι στη ρίζα τη επίλυση τη σύγκρουση. Δεν μιλάμε μόνο για κάτι ιδεαλιστικό, που αποτελεί μόνο ε, εντύπωση και αντίληψη της δύση. Όχι, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ βασικό για την σταθερότητα και την ε, ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Τρεις προκλήσεις λοιπόν ανέφερα ότι υπάρχουν. Να σας πω ποιες είναι. Καταρχάς, την ε, εξετάσει την πρώτη πρόκληση, το σημερινό φόρουμ. Το θέμα της συνοχής και της συνέπειας. Να σας πω ότι Πέρα από την πρόκληση της εξωτερικής και της εσωτερικής συνοχής σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων, υπάρχουν και άλλα δύο θέματα, η εξωτερική συνοχή και η εσωτερική συνοχή και οι σχετικές προκλήσεις που ανακύπτουν. Να σας πω τι εννοώ. Ε, εσωτερική-εξωτερική πρόκληση. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι όταν επισκεπτόμαστε χώρες σε όλο τον κόσμο και μιλάμε με οργανώσεις, με κυβερνήσεις και ζητούμε να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να περιμένουμε ότι πολλές, πολλές χώρες θα μας πούν, για παράδειγμα, «Α, και εσείς τι κάνετε με τους Ρωμά, με την ξενοφοβία» με τα εγκλήματα, τα ρατσιστικά στις χώρες σας, με τα οικονομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Πώς τα προστατεύετε αυτά σε μια εποχή κρίσης και ούτω καθεξής. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ερωτήματα και έγκυρα. Ω μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από κάποια χρόνια είχε συσταθεί μια ειδική επιτροπή η οποία εξέταζε κατά πόσον τα κράτη-μέλη ήταν νομιμιγμένοι και σε τι βαθμό στι παράνομε Απαγωγέ και στα βασανιστήρια των ε, περίφημων πτήσεων τη CIA. Αυτό αποτέλεσε μια αναγνώριση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο ότι κανείς δεν είναι τέλειος. Συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν θέλουμε να έχουμε αξιοπιστία και κύρος μιλώντα στο εξωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να το κάνουμε το ίδιο και στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανεί δεν είναι τέλειος, λοιπόν, αλλά μην με παρανοήσετε. Δεν εννοώ με αυτό ότι επειδή κανεί δεν είναι τέλειος, είμαστε όλοι εξίσου ατελεί στον κόσμο. Όχι, προφανώ και όχι και είμαι πάρα πολύ περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το, σε ενδεχομένω και των παραβιάσεων. Τρία κοινοβούλια έχουμε, συγγνώμη, έχουμε ελεύθερα κοινοβούλια όπου ο κόσμος έχει ελευθερία έκφρασης της γνώμης του, ελευθερία τύπου, ε, δημοσιογράφους οι οποίοι μπορούν να πούν ό,τι θέλουν χωρίς να φοβούνται ότι θα τους φυλακίσει κανείς έχουμε ε, και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε σωστούς υπαλλήλους. Έχουμε ε, μηχανισμούς οι οποίοι παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε τέλειοι δεν επιτρέπουν σε αυτές τις ατέλειες να λάβουν διαστάσεις όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. Τώρα, στη συζήτηση αυτή για την ιστορική, εξωτερική συνέπεια, τα κράτη-μέλη παίζουν σημαντικό ρόλο. Κάποια από τα θέματα που αναφέραμε, η ξενοφοβία, τα ρατσιστικά εγκλήματα, τα θέματα που αφορούν τον Ρωμά, όλα αυτά τα θέματα δεν είναι πάντα σε κάθε περίπτωση πανευρωπαϊκά προβλήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν πιο συχνά σε κάποια κράτη-μέλη από ό,τι σε άλλα. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας καλώ ως μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων να επαγρυπνείτε και για αυτά τα θέματα. Όχι απλά επειδή είναι σημαντικό για τα κράτη σας να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας, αλλά και γιατί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κάθε ένα από τα κράτη-μέλη είναι ένας πρέσβης, αν θέλετε, προς τον υπόλοιπο κόσμο των ευρωπαϊκών αξιών, των ευρωπαϊκών ανθρωπινών δικαιωμάτων. Αν στην αλυσίδα αυτή ένας κρίκος σπάσει, αυτό αποτελεί πρόβλημα για όλους. Δεύτερο θέμα που αφορά την συνέπεια. Εξωτερική, εξωτερική, εξωτερική, διπλά εξωτερική αν θέλετε, συνέπεια. Από έξω προς τα έξω. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αντιμετωπίζουμε κάθε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, μια παραβίαση ε, στην α χώρα καταδικάζεται εξίσου άμεσα όπως μια παραβίαση στην Β' χώρα, τρίτη χώρα πάντα. Ή μήπως έχουμε κάποιες προτιμήσεις ή θεωρείτε ότι έχουμε κάποιες προτιμήσεις σε κάποιες περιπτώσεις και αν θεωρείτε ή κάζετε ότι σε κάποιες περιπτώσεις κλείνουμε τα μάτια για παράδειγμα αυτό μήπως υπονομεύει από μόνο του τα, την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Εγώ θα σας πω ότι δεν αντιδρούμε πάντα με ακριβώς τον ίδιο τρόπο σε κάθε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητος απόρρια, αν θέλετε, σκοτεινών, ε, μακιαβέλιανών ε, σκέψεων και συμφερόντων. Αλλά να σας εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό. Πρέπει να το εξηγούμε αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται ίσως ε, για κάποια χώρα η οποία είναι πιο φιλική προς εμάς, προς κάποιο κρατός μέλος και αυτή η χώρα διαπράττει την παραβίαση. Και στην ε, περίπτωση αυτή καταλαβαίνουμε ότι ενδεχομένω να μην είναι ενδημικό και συστημικό το ζήτημα και μπορεί να χρησιμοποιούμε πιο ήπια διπλωματία λιγότερο δημόσια. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να θεωρούμε ότι δεν έχουμε ιδιαίτερη μόχλευση επί της χώρας η οποία διαπράττει την παραβίαση. Δεν υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, δεν υπάρχει τόσο, μεγάλη, ε, τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από πλευρά της χώρας για το δημόσιο ε, image της. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να πρόκειται για μια χώρα της γειτονίας μας, οπότε μπορεί να υπάρχουν πολλά οικονομικά, για παράδειγμα πολιτικά μέσα άσκησης πίεσης. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά αυτή την εξωτερική διάσταση της συνέπειας. Δεν είναι πάντα όμως, αν θέλετε, ένα θέμα ε, σκοτεινό. Τώρα, να μιλήσω, συνάδελφοι, για το θέμα της εσωτερικής συνέπειας. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό. Ανακύπτει το ερώτημα. Όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τα κράτη-μέλη, όλοι μας έχουμε ένα μήνυμα όταν μιλούμε για τις ε, χώρες και τα κράτη τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε συνεπείς μεταξύ μας ή μήπω επισκέπτομαι μια χώρα, καταδεικνύω κάποια θέματα και επισημαίνω κάποια θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά στη συνέχεια έρχεται ένας άλλος υπάλληλος ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάποια Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής, μεταβαίνει στην ίδια χώρα και έρχεται και λέει «Α, το ξέρω, ήρθε αυτός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά εμείς θα συζητήσουμε τώρα τα οικονομικά». Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για μία πρόκληση και πάλι δεν υπάρχει κακή, δεν υπάρχει πάντα δόλος, αλλά αυτό που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε πέρα από την μεγάλη επιτυχία του στρατηγικού πλαισίου που θα πρέπει να προωθηθεί σε κάθε διάσταση, στην περιβαλλοντική, στην εμπορική, πολιτική, κατά της τρομοκρατίας, σε όλα τα επίπεδα. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δεν είναι απλό. Δεν ασχολούνται όλοι με τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέκαθεν και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντική και αυτή η διαδικασία εσωτερικά. Σε αυτή την εσωτερική διάσταση είμαστε συνεπείς σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με πολυμερείς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και χαίρομαι ιδιαίτερως που παρευρίσκεται εδώ σήμερα με τα Ηνωμένα Έθνη, με τα περιφερειακά σώματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα προσπαθούμε να συνεργαστούμε μαζί τους προκειμένου να μην εμφανιζόμαστε απλά ως μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υποκρίνεται ότι είναι καλύτερη από τους άλλους, υποκρίνεται ότι έχει μαγικές λύσεις. Μπορούμε μαζί να βρούμε τον δρόμο για να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και επισημαίνω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα θα πρέπει να λέμε ακριβώς τα ίδια σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένω κάποιος να ακούγεται πιο πολύ και κάποιος ασκεί πιο ήπια παρασκηνιακή διπλωματία. Κάποιοι άλλοι παρεμβαίνουν σε διεθνείς οργανισμούς όπου έχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία. Αλλά να διαβάζουμε και να λέμε περίπου χοντρικά τα ίδια, να προωθούμε τους ίδιους στόχους σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδάλλως έχουμε εσωτερικά, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πρόβλημα. Δεύτερη πρόκληση λοιπόν πέρα από την συνέπεια. Πολύ σημαντικό αυτό γιατί έχει να κάνει για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και προκειμένου να μπορούν να εφαρμοστούν αποδοτικά θα πρέπει να καταστούν ιδιοκτησία του λαού σε κάθε χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υπόκειται πιέσεις αλλά τέλικη επιτυχία θα καθοριστεί κατά πόσο υπάρχει διεκτησία στο εσωτερικό της χώρας. Ε, κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών σε όλο τον κόσμο σήμερα δέχεται επιθέσεις. Με καταφανείς ε, τρόπους, ε, συγκίνονται συλλήψεις, φυλακίσεις εκτελέσεις ακόμα, αλλά και με πιο ήπιους, ύπουλους ε, τρόπους, ε, για παράδειγμα περιορισμός ε, της λειτουργίας των οργανώσεων. παρεμπόδιση της άσκησης του έργου αυτού των οργανώσεων και του λοιπά. Η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να έχει ένα χώρο ο οποίος θα προασπίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει να υπάρχει μια, μια ολοκληρωμένη προσήγηση. Κάθε φορά που πηγαίνουμε σε μια χώρα θα πρέπει να είμαστε πάντα σε επαφή με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Και εάν δεν είναι κίνδυνο, πηγή κινδύνου για αυτούς, να τους συναντάμε δημόσια. Πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους και πολλές φορές το κάνουμε πάρα πολύ αποτελεσματικά. Όταν λέω εμείς, ενώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Όταν παρακολουθούμε τις δίκες των αγωνιστών για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορεί να το κάνει μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία από τις πρεσβεία σας δεν μπορεί να το κάνει μόνη της. Αν συνεργαζόμαστε μπορούμε να το κάνουμε κάθε μέρα, να ξέρει το σύστημα σε κάθε χώρα ότι παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Θα πρέπει να δώσουμε χρηματοδότηση και δημιουργία, οικονομ... Ε, δημιουργία ικανότητας που είναι πιο σημαντική για την κοινωνία των πολιτών από ότι και τα χρήματα πολλές φορές. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κοινωνία των πολιτών και εμεί και σε όλο τον κόσμο και στις χώρες μας μπορούν να είναι ευγενικοί εάν το θέλουν, αλλά δεν χρειάζεται να είναι ευγενικοί έναντι των κυβερνήσεων. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να παρακολουθούν την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εφαρμογή της. Να παρακολουθούν και να καταγγέλνουν τις παραβιάσεις, να πληροφορούν τους ανθρώπους για τα δικαιώματά τους, να τους προστατεύουν πολλές φορές. Να προωθήσουν τη δημιουργία νομοθεσίας που να υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να δεχτεί όλα αυτά που της λένε οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Σημαίνει όμως αυτό ότι κάθε κυβέρνηση έχει μια απόλυτη υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι οι ΜΚΟ μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα χωρίς τρομοκράτηση και φόβο και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Και πάλι τα κράτη-μέλη μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο, εάν οι πρέσβοι σας και οι αντιπροσωπεία σας δεν συναντούν την κοινωνία των πολιτών στις χώρες αυτές, τότε έχουμε ένα πρόβλημα. Η τελευταία πρόκληση και εδώ θα κλείσω. Έχουμε την εξής πρόκληση που είναι διαφορετική. Τρία λεπτά, τέσσερα λεπτά. Η τελευταία λοιπόν πρόκληση. Αυτή δεν είναι μονάχα μια ευρωπαϊκή πρόκληση. Είναι μια παγκόσμια πρόκληση. Δεν είναι μονάχα μια πρόκληση που αφορά συγκεκριμένε χώρε όπω τα θέματα τη κοινωνία των πολιτών. Είναι μια θεμελιώδη πρόκληση για το υπόβαθρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι η επίθεση κατά τη οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βλέπουμε σε τόσο πολλέ περιπτώσει σε όλο τον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο ανέρχεται συνέχεια και ε, απλώνεται περισσότερο και υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα κατασκεύασμα της δυτικής κοινωνίας. Επομένως για να γίνουν δεκτά όλα αυτά στην κοινωνία μου θα πρέπει να γίνουν κοινωνικά και πολιτιστικά αποδεκτά στη δική μου κοινωνία και αυτό είναι δύσκολο και χρειάζεται χρόνο γιατί έχουμε τις παραδοσιακές μας αξίες οι οποίες πρέπει να τύχουν σεβασμού, θρησκευτικέ ή οικογενειακές αξίες οι οποίες αποκλίνουν από αυτά που λένε τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα. Αν αυτά τα επιχειρήματα επικρατήσουν και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουμε μάχες για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στάση σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη όταν πρόκειται για τη βία κατά των γυναικών. Και το Μάρτιο φέτος υπήρξε μια σειρά χωρών που προσπάθησαν να εμποδίσουν τα συμπεράσματα των ΗΠΑ για την καταδίκη της βίας κατά των γυναικών θέλοντας να τονίσουν περισσότερο τις οικογένειες αξίες. Αυτό το ξεπεράσαμε μια σημαντική μάχη. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει όλα τα κράτη-μέλη και ο κάθε κοινοβουλευτικό στις ε, χώρες μας να κάνει, να αγωνιστεί για τα θέματα αυτά. Πιστεύω πάρα πολύ στεναρά ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ήταν μια, μια μάχη μεταξύ θρησκειών ή μεταξύ πολιτισμών. Μια μάχη μεταξύ χωρών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν η παγκόσμια γλώσσα των φτωχών, των αδύναμων σε κάθε θρησκεία, σε κάθε χώρα, σε κάθε εθνικότητα εναντίον του σχετικισμού που ακολουθούν οι ισχυροί. Ποτέ δεν θα ακούσετε ένα θύμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να πει μην παρέμβετε να με βοηθήσετε γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι οικουμενικά. Πάντα θα ακούσετε όμως ισχυρούς τις κυβερνήσεις ότι δεν έχετε το δικαίωμα να παρέμβετε γιατί έχω παραδοσιακές αξίες. Ποτέ θα ακούσετε μια γυναίκα η οποία ξυλοκοπείται από τον άνδρα της σε κάποια χώρα του κόσμου, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας πει μη με βοηθήσετε γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι οικουμενικά. Είναι πάντα οι σύζυγοι, οι ισχυροί που θα πούν οι, οικο, οικογενειακές μου αξίες μου επιτρέπουν και μου επιβάλλουν να το κάνω αυτό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η η γλώσσα και οι αξίες των αδυνάτων, των ασθενών και όχι η γλώσσα των ισχυρών. Η κίνηση κατά της απεικιοκρατίας, οι επαναστατικές κινήσεις κατά της δύση ήταν ε, κινήσεις που διαπνεώτησαν με την ίδια γλώσσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τώρα ορισμένοι που καταπιέζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούν ότι πρέπει να χαρακτηρίσουν ως σχετικιστικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας και προσβλέπω σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας. Thank you. Ευχαριστούμε πάρα ε. πολύ για ε, την ένθερμη σου ε, ομιλία να αρχίσει τώρα η συζήτηση, να δώσω το λόγο σε όσους συναδέλφους είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια θέλουν να πάρουν το λόγο. Απλώς παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι σας, ίσως χρειάζεστε λίγο περισσότερο χρόνο για να το αποφασίσετε, αλλά σας ενθαρρύνω να πάρετε το λόγο. Και όσο καταρτίζεται ο κατάλογος των ομιλητών, ο πρέσβης Ρόισινς από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κύριος ε, Μπρόκ ε, είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα όταν συνέδεσε την Real Politik με τα ανθρώπινα δικαιώματα μας έχει δείξει, νομίζω, η ιστορία ότι δεν υπάρχει πραγματική ασφάλεια χωρίς ε, την, ε, τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μερικές φορές ε, ο κόσμος προσπαθεί να δημιουργήσει μία αντίφαση μεταξύ των δύο. Νομίζω όμως ότι κάθε φορά που υπάρχουν προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχει ε, και ένα, ένα αίσθημα έλλειψης ασφάλειας ε, ε, διεθνώς και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και σήμερα. νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των λαών συμμετέχουν σε αυτήν την διαδικασία και χαίρομαι ιδιαίτερα που συγκλήθηκε η σημερινή συνεδρίαση. Μια και βρίσκομαι ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σήμερα, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ψήφισμα τη κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη, το περασμένο φθινόπωρο, μετά από την εφαρμογή τη στρατηγική και του σχεδίου δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το ψήφισμα, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη εξέφρασε την ισχυρή τη ισχυρή υποστήριξη για τη δράση που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρει ειδικότερα τη σημαντική συνεισφορά των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γι' αυτό ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που καλωσορίζουμε σήμερα τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είπε ο ειδικό εντεταλμένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο κύριος Λαμπρινίδης, είναι πάρα πολύ στενές ε, και από την έγκριση του Μνημονίου Κατανόησης ε, από το 2007 μεταξύ των δύο οργανισμών βλέπουμε θετικές εξελίξεις. Ε, ήταν και ουσιαστικός στόχο του Γενικού Γραμματέα και των επικεφαλής των ευρωπαϊκών οργάνων. Έχουμε πολύ ε, πάρα πολύ καλές επαφές ε, στο ε, υψηλότερο επίπεδο και, και αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Οι νέες πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει νομίζουμε ότι αντικατοπτρίζουν μια νέα εποχή συνεργασίας ε, μεταξύ των δύο οργανισμών για την επίτευξη των κοινών μας στόχων. Αυτό έχει υλοποιηθεί με πολύ συγκεκριμένες ε, ε, περιπτώσεις. Τρία παραδείγματα θα αναφέρω. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει αυξανόμενο ενδιαφέρον και αυξανόμενη υποστήριξη για την επικύρωση σημαντικών συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης είτε μέσω των κρατών μελών, είτε από τα κράτη-μέλη της, ε, είτε από άλλα ε, ε, μέλη στα οποία εστιάζει την εξωτερική της πολιτική. Ενθαρρύνει την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω νομικώς δεσμευτικών κειμένων. Και αυτό ισχύει κυρίως για, το, για τη σύμβαση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο της Βουδαπέστης, ε, τη σύμβαση κατά της ε, ενδοοικογενειακής βίας, ε, της προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την σύμβαση Λαντζαρότο, όπως επίσης και την σύμβαση σώματεμπορίας κατά της σωματεμπορίας, ε, με την ε, υποστήριξη της επικύρωσης αυτών των ε, νομικών μέσων, είτε μέσω της προσπάθειας του κυρίου Λαμπρινίδη, είτε μέσω άλλων φορέων, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει μέσω καινοτόμων μέσων που βοηθούν την ενίσχυση των αξιών που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πρώτον, προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κάτι που υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τα Εθνικά Κοινοβούλια και είναι μια ορατή ένδειξη της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρεί στη Σύμβαση για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση της προσχώρησης ε, κάθε νομική πράξη της πρέπει να σέβεται τις διατάξεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα διαφορετικά ε, θα υπόκειται στην ε, ε, παρακολούθηση από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Οι δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί και ενώπιον του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι σημαντικές ε, σημεία αναφοράς για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συχνά υπάρχει συχνή συνεργασία μεταξύ ειδικών φορέων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μέσω της ε, Επιτροπής της Βιέννης, όπως επίσης και του φορέα που ασχολείται με την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων. Εμείς συμφωνούμε απολύτως ε, με την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεργασία με τους φορείς του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, μέσω επαφών σε υψηλό επίπεδο και αμοιβαία συνεργασίας. Βλέπουμε στην πράξη πολλά παραδείγματα επικοδομητικής συνεργασίας. Ε, αυτό βέβαια οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη δουλειά του κυρίου Λαμπρινίδη, του ειδικού εντεταλμένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον οποίο υποστηρίζω πλήρως γιατί είναι η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν διατρανώνει την, ε, την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης πιστεύουμε ότι τέτοια ενισχυμένη συνεργασία με τους ειδικού φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι χρήσιμη ε, στην επίτευξη ε, των νέων, και των νέων πρωτοβουλίων που έχουν αναλυφθεί για την παρακολούθηση της εφαρμογής ε, της στρατηγικής. Έχουμε παρακολουθήσει σε μεγάλο βαθμό την την επιστολή που απεστάλλει ε, προς τον ε, ε, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Παρόσο και τις σχετικές απαντήσεις που έδωσε στην, πρόσφατη ομιλία του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέλος της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Λουί Μισελ αναφέρθηκε σχετικά και στην έκθεσή του παρουσία στην Ολομέλεια του Στρασβούργου πριν από λίγες εβδομάδες. Επίσης ε, τονίζουμε ότι είναι πολύ ε, σημαντικό να ε, μην γίνεται διπλή δουλειά. Ένα σύστημα ανάπτυξης δικτών, παρακολούθησης και ανάπτυξης συστάσεων υπάρχει ήδη όπως γνωρίζετε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε λοιπόν οποιοδήποτε μελλοντικό μηχανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει υπόψη υπάρχοντες φορείς παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης στα οποίους έχουν προσχωρήσει καθορίσει όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόκειται για διεθνή μέσα τα οποία είναι ε, εξίσου νομικώς δεσμευτικά για όλα τα μέλη του Συμβουλίου ε, και πρόκειται για μη πολιτικοποιημένη αξιολόγηση, καθοδήγηση και μερικές φορές πρακτική συνεργασία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και έχουμε δει πολλά τέτοιου είδους παραδείγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρέσβη. Και τώρα έχουμε του κύριε Χαβέκβιν Αλτόντο από το Ισπανικό Κογκρέσο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ομιλώ εξ ονόματο του Ισπανικού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σύγκληση αυτής της συνεδρίασης και το Σταύρο Λαμπρινίδη για την παρουσία του σε αυτήν την ε, διοργάνωση αλλά και γενικά για το έργο του. Θα ήθελα όμως να αναφέρω και ένα τέταρτο στόχο, εάν αυτό είναι δυνατό, για το στρατηγικό σχέδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με ένα σημαντικό παίκτη στη ζωή μας. Δεν είναι πρόβλημα μονάχα οι κυβερνήσει. δεν είναι μονάχα η κοινωνία των πολιτών που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα θέματα ανθρωπινών δικαιωμάτων. Υπάρχει και ένας ακόμα σημαντικός εταίρος στην παγκόσμια οικονομία που είναι οι επιχειρήσεις. Όλο και περισσότερο στον χώρο δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που έχουν πολυεθνική προβολή και εργάζονται σε όλα τα τμήματα του κόσμου, λαμβάνουν χώρα παραβιάσεις ή καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είτε οι παραβιάσεις αυτές είναι στον κοινωνικο-οικονομικό τομέα είτε σε ένα ευρύτερο χώρο, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια τεράστια λυσίδα προβλημάτων που συνδέονται με την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Εγώ, ε, Σταύρο, έχω εκπλαγεί για το γεγονός ότι μέσα στο έργο μας, μέσα στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουμε συμπεριλάβει την αναζήτηση της, ε, εφαρμογής των αρχών του Ράγι. Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες, ε, τα Ηνωμένα Έθνη, συγγνώμη, έχουν δημιουργήσει ένα νέο εργαλείο που είναι η δημιουργία τριών βασικών αρχών που έχουν να κάνουν με τις κυβερνήσεις, με τις επιχειρήσεις και με τη δικαστική εξουσία όλων των χωρών του κόσμου, ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να καταγγείλουμε τις παραβιάσεις της παραβίας Οι επιχειρήσεις που έχουν εξορυκτική δραστηριότητα, κλωστοεφαντουργικά, εταιρείε μεταφορών, όλες αυτές οι εταιρείε έχουν να μας δείξουν μια προβληματική όλο και πιο πολύπλοκη σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ο Ράγκη στα, Ηνωμένα Έθνη μας έδωσε μια δυνατότητα να έχουμε ένα κοινό κώδικα, ένα οικουμενικό κώδικα, ένα ελάχιστο επίπεδο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε όπως είπε ο Σταύρος, τα ανθρώπινα δικαιώματα να γίνουν πια ένα παγκόσμιο νομικό και εκτιμένο, να είναι ένας κανόνας που να εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα του κόσμου, πέραν των εθνικών παραδόσεων, πέραν των νομικών διατάξεων της κάθε χώρας. Και αν η επιχείρηση δεν τηρεί αυτούς τους κανόνες θα μπορεί να τύχει καταγγελίες συντρόφισσες και σύντροφοι. Θέλω να σας υπενθυμίσω το πρόβλημα αυτό το οποίο έχει γίνει πριν από έξι μήνες στο Μπαγκλαντές με τις κλωστοϊφαντουργικές εταιρείε. Αν αυτές οι εταιρείε, οι ευρωπαϊκές και οι αμερικανικές που λειτουργούσαν στο Μπαγκλαντές σε ένα χώρο, σε ένα βιομηχανικό χώρο που μετά από την πυρκαγιά οδήγησε στο θάνατο 1.500 ατόμων και τραυματισμό πολύ περισσότερων ατόμων Αν είχαν καταγγελθεί στα ε, δικαστήρια της Νέας Υόρκης του Λονδίνου ή της Μαδρίτης με τον τρόπο, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν <clears throat> παραβιάζοντας απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εάν είχαν καταγγελθεί στα εθνικά δικαστήρια των χωρών αυτών, θα είχαμε κάνει ένα τεράστιο άλμα στην εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό, αγαπητέ Στάδο η δική μου πρόταση είναι, και η οποία προέρχεται και από το Ισπανικό Κοινοβούλιο, το οποίο πριν από λίγους μήνες μονάχα ενέκρινε μια τέτοια απόφαση, είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται με απόλυτο τρόπο και πλήρως οι αρχές ράγκη στην ε, ε, υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Ισπανία υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα είναι γιατί δεν κάνουμε τα απαραίτητα ώστε οι αρχές αυτές των Ηνωμένων Εθνών να είναι και έμπνευση για πολιτικές <clears throat> ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες και να αναφέρονται ιδίως στις ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις όταν λειτουργούν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τηρούν μέχρι και στα ανθρώπινα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές τις αρχές. Γιατί με τον τρόπο αυτό εμείς ως Ευρωπαίοι θα μπορέσουμε να κάνουμε σαφές τι είμαστε και τι θέλουμε να κάνουμε σε σχέση με το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας διαβεβαιώσω ότι στο Κοινοβούλιο είχαμε δύο α, εκθέσεις για, τα, για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το παρακολουθούμε το θέμα και σε ό,τι αφορά τον ΟΗΕ και τις συστάσεις του. Αυτά είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά για μας. Συχνά γίνονται λοιπόν συζητήσεις για την ενδυνάμωση των συστάσεων του ΟΗΕ, γιατί φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι πρόβλημα το γεγονός ότι δεν είναι για πολλές επιτροπές νομικά δεσμευτικά οι συστάσεις αυτές. Επίσης ασχολούμαστε με θέματα διαφθοράς και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάλι εστιαζόμαστε στο συγκεκριμένο ρόλο των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μεμονωμένες χώρες. Δύο μιλητές έχω από τα Εθνικά Κοινοβούλια και μετά θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις από τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγγνώμη τώρα, έχουμε τον ε, κύριο Ντόνσκι από τους ε, Λιθουανία και από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, πολλά σημαντικά θέματα ανέφερε στο Λαμπρινίδης και τον χαιρετίζω και τον συγχαίρω για την εξαιρετική του δουλειά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ακριβής, ενδελεχής στη δουλειά του. Και ήταν πραγματικά μεγάλη παρέμβαση στη συζήτησή μας. Θα ήθελα λοιπόν Σταύρο να, να συγχαρώ για την ολιστική σου προσέγγιση, για την έμφαση που δίνει στον κρίσιμο ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη σταθερότητα και την ειρήνη στον κόσμο. Αντί να δώσεις μια ιδεαλιστική διάσταση στα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο δεν ισχύει στον κόσμο που ζούμε. Χάρηκα λοιπόν που έδωσες έμφαση στην κοινωνία των πολιτών, στις ΜΚΟ και θα ήθελα να σου επιστήσω την προσοχή στο εξή σε διαφορά μεταξύ των πραγματικών ΜΚΟ που καταγράφουν την ε, κατάσταση σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες και στον κόσμο, αλλά μεταξύ αυτών των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των άλλων που έχουν, αν θέλετε, εξημερωθεί και έχουν, ε, εξυπηρετούν συμφέροντα. Και αυτό συμβαίνει σε πολλές ε, χώρες όπου υπάρχουν ΜΚΟ που θεωρούμε ότι είναι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ουσιαστικά εξυπηρετούν συμφέροντα. Θα πρέπει λοιπόν να τις διακρίνουμε αυτές τις οργανώσεις από αυτές που πραγματικά δραστηριοποιούνται. Κάτι άλλο, και το έχουμε συζητήσει αυτό σε πολλές περιστάσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιστοί στις θέσεις μας σε ό,τι αφορά την ανάγκη να υποστηρίξουμε τους ακτιβιστές και τους προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους αντιφρονούνται σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς. Θα πρέπει όχι μόνο να τους σεβόμαστε, αλλά και να τους προστατεύουμε γιατί οι Κινέζοι, οι Ρώσοι αντιφρονούντες είναι οι πιο πολύτιμοι σε ό,τι αφορά την πολιτική του ουσία σε όλο τον κόσμο. Είναι κρίσιμη σημασία η προστασία τους και νομίζω ότι χρειάζεται πιο πολύ συνεργασία από πλευρά μα με κέντρα, με δημόσιες οργανώσεις που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε συνεργασία με συγγραφείς, με ενώσεις. Και τέλος, είναι πολύ σημαντικό να το επαναλαμβάνουμε διαρκώς ότι η πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αποτελεί άδεια να είναι κανείς επιλεκτικός συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών όπου υπάρχουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί πολλά δημοκρατικά κράτη κάνουν παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ούτε είναι αυτό δικαιολογία για να επιτιθόμεθα σε χώρε που δεν μα αρέσουν. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια καθολική παγκόσμια γλώσσα που μα επιτρέπει να κατανομάζουμε και να δακτυλοδεικτούμε τι χώρε εκείνες που θέλουν να προσπίζονται με τα δικαιώματα αλλά δεν σέβονται τους πολίτες τους. Ευχαριστώ κυρία Ντότσκης, η κυρία Χριστίνα Τιπιέτρο από την Ιταλική Γερουσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μια μεγάλη χαρά να είμαι εδώ και να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ένα θέμα που είναι τόσο σημαντικό και το οποίο όλο και περισσότερο το αντιλαμβάνονται η Εθνική Κοινοβουλευτική και η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική ως μία προτεραιότητα. Η κίνηση πέντε αστέρια στο εσωτερικό της Ιταλικής ε, Γερουσίας βλέπει με πολύ θετικό μάτι την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της προτεραιότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μεγάλη λοιπόν προσοχή έχουμε παρακολουθήσει την πρόταση που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πακέτο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το πολύπλοκο αυτό θέμα το οποίο οξύνεται ιδιαίτερα με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που έχει δείξει όλα τα κράτη-μέλη και που απαιτεί μια κοινή προσπάθεια για να γεφυρωθεί το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των θεσμών και των πολιτών. Είναι απαραίτητο λοιπόν σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό να υπάρξουν συνέργειε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στα καλύτερα αποτελέσματα. Μια βέλτιστη δράση για, τη, για το στρατηγικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθώντα τι κατευθυντήρε γραμμέ του σχεδίου δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Είναι λοιπόν επιτακτικό για όλους μας να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις που έχει ενώπιον της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη δική μας άποψη το να μπορέσουμε να μετατρέψουμε αυτές τις αρχές σε συγκεκριμένες δράσεις, να είμαστε λοιπόν στο κέντρο αυτών των προβληματικών και να ξεπεράσουμε το να είμαστε απλώς μια ακαδημαϊκή άσκηση και να προχωρήσουμε σε δράσεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα που θίγουν ένα πολύ μεγάλο μέρος ατόμων που είναι ευάλωτα λόγω της κοινωνικής προέλευσης, όλο αυτό πρέπει να είναι ένα εγχείρημα το οποίο θα πρέπει να διέπεται από πραγματισμό. Οι γραμμές που αναφέρουν το σχέδιο δράσης, δηλαδή η ανάπτυξη εθνικών σχέδιων για την δράση, ώστε να εφαρμοστούν αυτές οι αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να γίνει με το να δοθούν όλες οι απαραίτητες υποστηρίξει σε δράσεις όπως αυτή που αναπτύσσει η Ιταλική κυβέρνηση μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσεως. Είναι απαραίτητο λοιπόν να βοηθήσουμε να ακολουθήσουν και τα άλλα κράτη θετικά παραδείγματα όπως αυτό της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Σας ευχαριστώ. Μας υπενθυμίσατε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι νομίζω το μοναδικό εθνικό κοινοβούλιο έχει το μοναδικό Εθνικό Κοινοβούλιο με ένα εθνικό σχέδιο δράση για τι επιχειρήσει και τα ανθρώπινα δικαιώματα ω τώρα. Τέλος, κλείνοντας, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Άννα Αλλά πού είναι, δεν τη βλέπω. Ίσως αργότερα να θέλει το λόγο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνουμε input και από τις ε, οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. Να ακούσουμε λοιπόν δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, από τις Βρυξέλλες, μετά τις Βρυξέλλες. Human Rights Watch, Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να λάβουμε το λόγο σε αυτή την πολύ σημαντική ακρόαση. Ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλες τέτοιες ακροάσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων ε, με σκοπό την αναζήτηση καλύτερων τρόπων εφαρμογής ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, παγκοσμίω. Εγώ συμφωνώ απολύτως ε, με όλα όσα υπόθηκαν από τον ειδικό, ε, τον ειδικό αντιτελμένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον Σταύρο Λαμπρινίδη. Νομίζω ότι σωστά μας είπε σε, ό, μας είπε σε όλους, μας υπενθύμησε ότι ήταν αποτέλεσμα τα ανθρώπινα δικαιώματα συλλογικής προσπάθειας που δεν θα είναι επιτυχής παρά μόνο αν υπάρξουν οργανωμένες προσπάθειες από τις κυβερνήσεις, από τα εθνικά κοινοβούλια ε, από την κοινωνία των πολιτών ε, και από την Ε.Ε. Υπάρχουν ε, διάφορα προβλήματα σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά φιλόδοξα αποτελέσματα καταφέραμε ε, την περασμένη χρονιά με επικοδομητική συνεργασία. Ο Σταύρος μας το υπενθύμησε και αυτό, ότι η επόμενη φάση είναι η δυσκολότερη, ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τώρα όλα αυτά που αποφασίσαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και χωρίς ε, συλλογική ε, ενθάρρυνση και πυγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα, δεν θα επιτύχουμε στο βαθμό που θα έπρεπε. Να σας δώσω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα του τι προτείνουμε εμείς για να ε, προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Δεν θα χρησιμοποιήσω τα πέντε λεπτά μου για να μιλήσω για τις, ε, όλες αυτές τις ωραίες αρχές και αξίες, αλλά για κάτι πολύ συγκεκριμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάντοτε εγκρίνει πολύ ε, σημαντικά και ισχυρά ε, ψηφίσματα, αλλά δεν θα μπορέσει να προωθήσει αυτό το ε, μήνυμα των ψηφισμάτων χωρίς τη βοήθεια των Εθνικών Κοινοβουλίων. Το στρατηγικό πλαίσιο και το πακέτο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι θα υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όλους όσους είναι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους στρατηγικούς εταίρους. Ελπίζω και η δοκιμή αυτή ε, της ε, προσπάθειας θα γίνει. Δηλαδή θα δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση πόσο υπέρμαχος είναι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τη Ρωσία και την Κίνα, δύο σημαντικούς στρατηγικούς εταίρους, αλλά επίσης και σοβαρούς παραβάτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Σταύρος πολύ σωστά είπε ότι όλοι πρέπει να ε, μιλούμε με μία ενιαία φωνή. Όμως ε, δεν έχει οριστεί απολύτως ε, αυτή η ενιαία φωνή γιατί η ΕΕΔ μιλά συχνά με διάφορες φωνές όσον αφορά διάφορα προβλήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας καλούμε και αυτό είναι κάτι που το ζήτησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από ένα χρόνο και στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλα ψηφίσματα ε, σας κάνουμε έκκληση μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς να έχουμε ε, ισχυρά αποτελέσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων με συγκεκριμένα μηνύματα, συγκεκριμένη συλλογική στρατηγική για το πώς θα ε, προαγάγουμε τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως ε, σε σχέση με τη Ρωσία και την Κίνα. Αυτό το μήνα ε, μέσω των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων υποθέσεων από τους υπουργούς εξωτερικών δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι ένας κοινό παρονομιστής. Δεν μπορεί κανείς να πάει να κάνει λιγότερα, μπορεί να κάνει περισσότερα, αλλά όχι λιγότερα. Δεν μπορεί κάποιος να έχει διάλογο με τη Ρωσία και την Κίνα και να μην εκπροσωπεί αυτό το συλλογικό μήνυμα. Άλλο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι μπορεί ε, κανείς ε, ε, να συλλογικά να προωθήσει κάτι πολύ καλύτερα από ό,τι μεμονωμένα είναι ένα μήνυμα, θα λέει ο κάθε εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, που είναι ένα τμήμα του μήνυματο της ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και καθένα ε, μπορεί να εκπροσωπήσει αυτό το μήνυμα, να το μεταφέρει έχοντα πίσω του την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι η Κίνα και η Ρωσία δεν μπορεί εύκολα να το αγνοήσει γιατί ε, δεν θα υπάρχει σοβαρή υποστήριξη, θα υπάρχει πίσω, από πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει ένα κοινό μήνυμα το οποίο θα προσπαθούν να το εκπροσωπούν όλοι. Δεν θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό αν δεν υπάρξει ενθάρρυνση, ενίσχυση από, το, ε, από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ελπίζω λοιπόν να... Ε, το αποτέλεσμα της σημερινή ακρόασης να είναι αυτό, ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια και εκείνα θα συμμετέχουν. Επίσης, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ε, και ενώπιον χωρών όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιο κύρος. Το Μπαχρέιν είναι μία από αυτές τις χώρες. Ε, στην Αραβική ε, Άνοιξη, το, λόγω της Αραβικής Άνοιξης, το Μπαχρέιν ε, επλήγει, βρίσκεται σε μετάβαση, αλλά θα έχει μπροστά, ένα δύσκολο έχει μπροστά του ένα δύσκολο ε, δρόμο. Στον Παχρέιν όσοι διαδήλωσαν στους δρόμους ζήτησαν ειρηνικά την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους ε, και επέκριναν ειρηνικά τα, ε, τις κυβερνήσεις τους, όμως πλήρωσαν ένα πάρα πολύ σοβαρό τίμημα και έχουν τώρα βρεθεί φυλακισμένοι αυτή η ειρηνική, ε, αυτό το ειρηνικό κίνημα ε, στο οποίο συμμετείχε και ένας ε, στο οποίο συμμετείχε και Ευρωπαίος πολίτης, ε, είχε ω αποτέλεσμα να βρεθεί ο άνθρωπος αυτός ε, στη φυλακή. Υπάρχουν άνθρωποι που ειρηνικά διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους, για πράγματα τα οποία εμείς έχουμε πει ότι θα υποστηρίξουμε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα βρίσκονται στι φυλακέ του Μπαχρέιν. Πρέπει να βρούμε ένα συλλογικό τρόπο εξασφάλισης ε, των ελευθεριών ανθρώπων που πληρώνουν πολύ μεγάλο τίμημα σήμερα. Ε, μερικοί έχουν ε, καταδικαστεί σε ισόβια κάθυρξη και ακόμα δεν έχουμε ένα ισχυρό μήνυμα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον από την ε, δεν υπάρξουν πιέσεις για να αλλάξει, δεν υπήρχαν πιέσεις για να αλλάξει κάτι δεν υπάρχουν μηνύματα συλλογικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να καθιστούν σαφές ότι αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να, είναι, ε, να βγει από τη φυλακή, να είναι μέσα στη φυλακή και, η κυβέρνηση του Μπαχρέιν πρέπει να ε, κάνει διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτό. Παρακαλώ ολοκληρώστε, παρεμβαίνει η Πρόεδρος. Μία τελευταία παρατήρηση και το λέω αυτό τώρα γιατί δεν είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσω να ξαναπάρω το λόγο μετά. Υπήρξε γενικώ ε, μία δυσαρέσκεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το δημοκρατικό έλλειμμα, τη, σε σχέση με τις ε, αποφάσεις που λαμβάζονται και στο τομέα των, ε, των εξωτερικών υποθέσεων ε, επειδή η απόφαση είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εκτελούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης κάτι το οποίο δεν είδε ποτέ κανένας Ευρωπαίος πολίτης ούτε η κοινωνία των πολιτών οι Υπουργοί Εξωτερικών να συζητούν μεταξύ τους. Δεν το έχουμε δει ποτέ αυτό. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας ζητήσω ετησίως ε, να γίνεται μία συζήτηση της, ε, για τη στρατηγική και το πακέτο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με, μεταξύ των, των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα δεσμεύονται και θα λένε ακριβώς τι θέλουν να επιτύχουν. Θα χρειαστεί να είμαι λίγο πιο αυστηρή με το χρόνο, λέει η Πρόεδρος, γιατί θα ήθελα να ακούσω και τις απαντήσεις του Σταύρου Λαμπρινίδη. Vincent Forrest από τους Frontline Defenders. Θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, είμαι από μια οργάνωση η οποία δεν είναι τόσο γνωστή σε σχέση με την Human Rights Watch, Frontline Defenders, η διεθνή ε, οργάνωση για την υπεράσπιση των πρόσπιστων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προηγούμενη εβδομάδα γιορτάσαμε την απελευθέρωση του βραβευμένου με το βραβείο Σαχάροφ το 2012. Όπως είπε και ο κύριος Ντόνσκιν και ο κύριος Λαμπρινίδης υπάρχει ανάγκη τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προασπιστούν αυτούς που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί αυτοί είναι οι πρωταθλητές, αυτοί είναι που διακυβεύουν τη ζωή τους και αυτοί μπαίνουν στο στόχαστρο γιατί προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και μόνο τρία σημεία του σχεδίου δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν να κάνουν με αυτού του προασπιστέ των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πρόκειται όμω για ένα εγκάρσιο ζήτημα. Σύμφωνο με τον κύριο Μπροκ και τα εισαγωγικά του σχόλια που μίλησε για κοινή ευθύνη. Το σχέδιο δράσης δεν είναι μόνο θέμα για την υπηρεσία εξωτερική δράση και την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου. Όχι. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί όλους, όλου τους εκπροσώπους και όλα τα κοινοβούλια, τα εθνικά κοινοβούλια τα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να σπρώξουν τι κυβερνήσει για να διαδραματίσουν το ρόλο που τους ερμόζει σε ό,τι αφορά τους προσπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, καταπήγοντα ψηφίσματα, επιστολές προς τις πρεσβείες, για συναντήσεις, αποστολές τόπου όπου μπορεί κανείς να συναντήσει τους ανεξάρτητους προσπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, να ακούσει ποιες είναι οι ανάγκες τους, στη συνεργασία με τις ΜΚΟ σε διεθνές και ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο και εθνικό επίπεδο συναντήσεις στις πρωτεύουσες και στις Βρυξέλλες. Στρατηγικές, ε, εταιρικέ ε, σχέσεις, ε, συμφωνίες. Θα ήθελα να κάνω και 7 επιπλέον συστάσεις, αν μου επιτρέπετε, όσο πιο πρακτικές γίνεται. Υπάρχει μια σαφή στάση μετά από την συνθήκη της Λισαβόνας να πούμε ότι α, εξαρτάται και είναι θέμα των αντιπροσωπείων να φροντίσουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πράσπιστές αυτών. Άρα, παρά το γεγονός ότι είναι τα σημεία επαφής σε κάθε, σε κάθε χώρα, έχουν ε, βάση στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία. Καλό και κακό. Γιατί? Γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια σημεία εστίασης στις πρεσβείας και θα πρέπει να υπάρχει κοινή ευθύνη και ιδιοκτησία. Κατά δεύτερον, να υπάρχουν συγκεκριμένα ψηφίσματα για τους πρασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη Γερμανία γίνεται αυτό και προσφάτως έγινε και στο Βέλγιο. Τρίτον, οι περικοπές στον προπολογισμό να μην επηρεάζουν τα προγράμματα το κυβερνητικά για την υποστήριξη των, ε, της των πολιτών. Κατά τέταρτον, να υπάρχει μία ε, πρωτοβουλία δραστηριο, ε, μία πρωτοβουλία αδελφοποίησης. Να εντοπίζονται ποιοι έχουν μπει στο στόχαστρο. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με προγράμματα ευρωπαϊκού και εθνικών κοινοβουλίων. Πέμπτον, θα πρέπει να εξετάσουμε τη δημιουργία ενός δικτύου κατεπίγουσας ανάγκης για να υπάρχει ταχεία ανταπόκριση. Όχι μόνο μέσω της διαδικασίας και της πρωτοβουλίας αδελφοποίησης. Και αυτό θα μπορούσε να υποστηρίξει τη ΣΜΚΙΟ. Έκτον, σύσταση στην ε, έκθεση τεράς ένα, για την οργάνωση της εκδήλωσης ε, στις Βρεξέλλες για τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Διαφορετικό διαφορετική εκδήλωση από το βραβείο Ζαχάροφ, με έντονη δημοσιότητα, με ένα ψήφισμα, συγκεκριμένε δραστηριότητε που θα διοργανώνονται, εκπαιδεύσει ενδεχομένω. Και τέλος, να σκεφτούμε λίγο πιο ευρέω. Κοινωνικά δίκτυα, για παράδειγμα, χρήση τοπικών μέσων ενημέρωσης στις εκάστοτες χώρες για να ακούει και η κοινή γνώμη τι γίνεται. Και όλο αυτό θα δώσει μια νόμιμη διάσταση στο έργο των πρόσπιστων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης να σας ενημερώσω ότι εμείς έχουμε δημοσιεύσει ένα εγχειρίδιο σε σχέση με το τι μπορεί να περιμένουν οι προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά και στο Ευρωπαϊκό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναφέρει και εσάς ω ευρωβουλευτέ. Σα ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για τι συστάσει σα, λέει ο Πρόεδρο, Σε ό,τι αφορά του προσπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήθελα να καλωσορίσω και μια αντιπροσωπεία από το Κοινοβούλιο της Μιανμάρ που παρακολουθεί την συζήτηση. Καλώ ορίσατε. Πρόκειται για μια συνεδρίαση μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μέλων, μέλων ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων που ασχολούνται με θέματα εξωτερικών υποθέσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πριν δώσω το λόγο στον Σταύρο Λαβρενίδη για κάποια καταληκτικά σχόλια, νομίζω ότι το δίκτυο των θεσμικών ε, οργάνων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πάρει το λόγο εν συντομία. Τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κριστόφερσεν, Είμαι επικεφαλής του Δανικού Ινστιτούτου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λειτουργεί. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Δείτε Κριστόφερσεν λοιπόν, από το Δανικό Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Δανία και, υποστηρίζω, και εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Ιδρύματα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που δημιουργήθηκε φέτος. Ένα από τα κύρια θέματα που μας απασχολούν στον εαυτό δίκτυο είναι συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πέρσι το 2012 εγκρίναμε τις λεγόμενες αρχές του Βελιγραδίου σε σχέση με τη συνεργασία Εθνικών Κοινοβουλίων και Εθνικών Ιδρυμάτων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι εσείς έχετε τα λάπτοψ και άμα κάνετε ένα γουγλάρισμα θα μπορείτε να βρείτε τις αρχές του Βελιγραδίου και να δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις αρχές για να έρθετε σε επαφή και να λειτουργήσετε με τους Εθνικούς Φορείς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο δικός μας στόχος για τη βοήθεια των ε, κοινοβουλίων είναι πολύ σημαντικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό έχουμε ένα γραφείο στις Βρυξέλλες για να είμαστε πιο κοντά στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο το Κοινοβούλιο, αλλά το Φορέα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το, την Κομισιόν κτλ. Ένα κύριο θέμα λοιπόν το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό αυτό δίκτυο είναι η απουσία πλήρως ανεξάρτητων Ιδρυμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα μονάχα υπάρχουν 12 κράτη-μέλη που έχουν Κατηγορία Α ιδρύματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενώ όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει άλλα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσουν τέτοιους θεσμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επικρατήσει πλήρως αυτό. Γιατί ζητάει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητά από τις χώρες που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν τέτοια Ινστιτούτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν δεν ισχύει αυτό για τα περισσότερα κράτη-μέλη. Για να είμαι λοιπόν σύντομο με στον χρόνο που μου έχει δοθεί, κυρία Πρόεδρε, απλώς μια κύρια αίτηση και πρόταση από το δίκτυο α, Ιδρυμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σας ζητώ όλους να εξετάσετε πώς μπορούν να δημιουργηθούν εθνικοί θεσμοί και να ενισχυθούν σε όλα τα κράτη-μέλη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σας ζητώ επίσης να εξετάσετε αν θα ήταν πολύ σημαντικό να εξασφαλίσετε την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και η Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και να εγκριθεί κάποιο νομοθέτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιβάλλει στα κρατη τη δημιουργία θεσμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να εφαρμόσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα <clears throat> στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της. Ευχαριστώ κύριε Κριστόφερσον. Σταύρο, υπάρχει ένα ερώτημα προς εσένα για από κάποιο μέρος ένα λεπτό μονάχα για να μπορέσει να, για να απαντήσει. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία ελέγχθηκαν σε αυτή την αίθουσα είναι η δυσκολία μιας κοινή εξωτερικής στάσης όταν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη δική μου εμπειρία υπάρχουν χώρες οι οποίες ακούνε πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία λέμε και αυτά τα οποία λένε τα διεθνή δικαστήρια τα οποία προσπαθούν να εξασφαλίσουν το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενώ άλλε χώρε δεν δίνουν κανένα, ε, καμία βάση, κανένα, καμία συνέχεια σε όλα αυτά τα θέματα και συνεχίζουν τι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρουμε ότι αυτή η έλλειψη προσοχή στα θέματα αυτά εξαρτάται από την πολιτική και οικονομική ε, εξουσία και δύναμη των χωρών αυτών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε πάντα ως Ευρωπαϊκή Ένωση να καλούμε τις χώρες αυτές να, να αντιμετωπίσουν και να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα ιδιαίτερα όμως να σταθώ στη θέση των γυναικών και των κοριτσιών που χρειάζονται μια προστασία σε, στις ένοπλες συγκρούσεις όπου οι βιασμοί γυναικών και κοριτσιών έχουν γίνει πολεμικό όπλο. Επίσης έχουμε καταδικάσει την, τον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων και τους ε, γάμους με το ζόρι που ασκούνται σε πάρα πολλές χώρες. Υπάρχει καταδίωξη πολλών γυναικών και γυναικείων οργανώσεων σε πολλές χώρες του κόσμου. Πρέπει οι αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πιέσουν για να μπορέσουν οι χώρες αυτές να δεσμευτούν για μια μεγαλύτερη προστασία των γυναικών και των κολλησιών που ζουν με σχεδόν απόλυτη αποστέρηση των δικαιωμάτων τους. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λαβρινίδη πώς θα μπορούσαν λοιπόν οι αποστολές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στις χώρες αυτές όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται και πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προστασία. Ευχαριστώ. Πέντε λεπτά έχετε το λόγο τώρα. Thanks, thanks. No, no more. I... Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω να χρειαστώ περισσότερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και θα χρειαστεί να φύγω. Ζητώ συγγνώμη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω πολύ γρήγορα σε κάποια από τα ερωτήματα. Είναι μια πραγματική πρόκληση. πρέπει να δούμε τι μοχλό πίεση έχει κανείς. Είναι κάτι που πρέπει πάντοτε να το διερευνά. Μπορεί να, σε μια χώρα να μην ενδιαφέρονται για τα λεφτά σου, αλλά ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τη διεθνή σου εικόνα. Μπορεί να μην ενδιαφέρεται ο κόσμος σε μια χώρα για τα δικά σου λεφτά, αλλά για τα λεφτά μιας, ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους. Και μιλάω για, όταν λέω τα λεφτά σου εννοώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε πάντως Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ε, ερχόμαστε σε επαφή σε μια, σε, με, μια χώρα, πρέπει να σκεφτόμαστε την πυγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν, κάποια, όταν ε, μπλεκόμαστε σε μια χώρα για οποιοδήποτε ιστορικό, οικονομικό, κοινωνικό λόγο, αυτή η χώρα πρέπει να επιβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα εξίσου όσο εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έτσι θα κάνουν τη διαφορά αν το κάνουν αυτό δεν μπορούμε εμείς να νύπτουμε τα σχήρες μας και να λέμε μία χώρα ή η αλλη ε, είπε το ένα ή το άλλο. Σε πολυμερές επίπεδο λοιπόν πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με μεγάλους παίκτες της οικονομικής ε, σκηνής του της συγκεκριμένης ε, χώρας. Το ίδιο ισχύει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, στο να, ότι είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε αυτήν την ε, συλλογική μας πυγμή. Η Επιτροπή της Βιέννης, για παράδειγμα, του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, μας, μας βοήθησε να λύσουμε τα προβλήματα με μια πολύ αμφίβολη μη κυβερνητική οργάνωση σε μια χώρα. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα ε, των επιχειρήσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μόλις ήρθα από την Κίνα. Η πρώτη συνάντηση που είχα στην Κίνα ήταν ε, μια πρώτη στρογγυλή τράπεζα για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προσπαθήσαμε και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών και των κινέζικων επιχειρήσεων, ε, ε, ακαδημαϊκοί, άνθρωποι που προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να καθίσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι. Οι άνθρωποι που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα, προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να το κάνουν καλύτερα και όταν πηγαίνουμε στην ίδια τρίτη χώρα και εμείς και η Κίνα να εξασφαλίζουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, μεταξύ των οποίων και τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν παραβιάζονται. Εμείς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτέλεσε έμπνευση. Ξέρω η έκθεση Χάουαρντ, ε, αναφέρεται και άλλη μία έκθεση ε, Και αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο τα κοινοβούλια μπορούν να ε, κάνουν τη διαφορά. Όπως είπε ο Έλμαρ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες. Έχει όμως ε, πολιτική δύναμη ε, και ε, στις χώρες σας νομίζω ότι μπορείτε να καθοδηγήσετε το διάλογο προς αυτή την κατεύθυνση και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργάνωσε την ακρόαση αυτή. Ήδη από τον Ιούνιο του 2013 εξέδωσε τρία σημειώματα καθοδήγησης ε, σε χώρες ε, ε, μιλάω για τις αρχές Ράγκη που είναι ε, ο εισηγητής για τα Ηνωμένα Έθνη για το θέμα αυτό. Πρώτον για πετρελαϊκές εταιρείες και εταιρείες εκμετάλλευσης αερίου, εταιρείες ε, πληροφορικής και εταιρείες προσωρινής απασχόλησης. Η Επιτροπή Επίσης εξέδωσε ένα εσωτερικό έγγραφο για το πώς οι, ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές όταν δραστηριοποιούνται εντός της Ευρώπης. Οι πρώτες τρεις λοιπόν κατευθυντήριες γραμμές ήταν για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εσωτερικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τι γίνεται εντός της Ένωσης. Δεν είναι δεσμευτικές για την ώρα ίσως, αλλά Χαίρομαι που ε, ασκείται πίεση επί των θεμάτων αυτών και ε, το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο και ευχαριστώ και το Ισπανικό Κοινοβούλιο που τοποθετήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς πρέπει να φύγω γιατί πρέπει να συνεχίσω τις εργασίες μου για την Κίνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτιμώ ιδιαίτερος τις παρεμβάσεις όλων και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λαμπρινίδη, λέει πρόεδρος. Ελπίζω να σας έδωσε κάποια τροφή για σκέψη ε, η σημερινή μας συνεδρίαση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε ε, μια ε, πολύ καλή φωνή σε διεθνή φόρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στο επόμενο θέμα για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διεθνή φόρα. Ο κύριος Τόιρμαν είναι εδώ. Θα του ζητήσω να έρθει εδώ στο Προεδρείο. Να εξηγήσω επίσης πώς προετοιμάζουμε στο Κοινοβούλιο τα, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΙΕ ή το, τη Συνεδρία Γενικής Συνέλευσης ε, στη Νέα Υόρκη. Είναι δύο, είναι δύο διαφορετικά όργανα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στο ευρύ κοινό αν είναι σημαντική αυτή η δουλειά ή όχι, αλλά σίγουρα χρειάζεται πολύ μεγάλη υποστήριξη ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν εκπροσωπείται στα διεθνή ε, φόρα. Πριν πάει, για παράδειγμα, στο, στη Γενέβη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει ε, στην Ολομέλη ένα ψήφισμα για τις προτεραιότητές μας με τη συγκεκριμένη σύνοδο που λαμβάνει η χώρα συνήθως το Μάρτιο στη Γενέβη. Και κατά την προετοιμασία Έχουμε πολύ στενές επαφές με την κοινωνία των πολιτών, όπως επίσης και με κράτη-μέλη, για να δούμε ποια είναι η δική τους ε, άποψη, ε, προσέγγιση κατά την παρακολούθηση των, ε, φορέων, των εργασιών των φορέων του ΟΗΕ και πώς μπορούν επίσης να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στη Γενέβη και στη Νέα Υόρκη για τα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, έχει τη δυνατότητα να ε, μιλήσει ενιαία. Τα κράτη-μέλη ε, μιλούν μεμονωμένα. Γι' αυτό ο ειδικό εντεταλμένος δεν έχει την εντολή από τα κράτη-μέλη να μιλήσει εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όμως ε, στο Συμβούλιο ΙΚΟΧΟΜ ε, ένα, μια ομάδα εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ε, Συμβουλίου. Προσπαθούν να δουν με ποιο τρόπο πρέπει να δρουν σε διεθνές επίπεδο. Είναι εδώ ο κύριος Τόιερμαν που είναι ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό και ε, ξέρει ε, πολλά για την διαδικασία λήψης αποφάσεων, ε, κάτι το οποίο έχει βέβαια βελτιωθεί. Νομίζω ότι υπάρχει τώρα δυνατότητα να έρχεστε σε επαφή στις Βρυξέλλες με συγκεκριμένους ανθρώπους για την βελτίωση της πολιτικής αυτής. Ε, δύο φορές πηγαίνω στην ΕΚΟΧΟΜ, ε, ε, οι διπλωμάτες που εκπροσωπούν τις διάφορες χώρες εκεί κατανοούν ότι είναι σημαντικό να φτάνουν σε μια ευρωπαϊκή θέση και να μην παραμένουν στις εθνικές προτεραιότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, νομίζουμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό για τη σημερινή μας ακρόαση και για τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακούσουμε για τη δουλειά της ΚΟΧΟΜ από τον κύριο Τόιερμαν, τον πρόεδρό της, ε, να σας πούμε και εμείς ε, να ε, μεταφερθεί στις ε, διάφορες πρωτεύουσες των κρατών μελών ε, πόσο σημαντική είναι αυτή η ενιαία τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διεθνή φόρα. Να σας δώσω τώρα το λόγο γιατί να μας πείτε περισσότερα πράγματα για τη δουλειά της ΚΟΧΟΜ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και μεγάλη μου τιμή που συμμετέχω σε αυτό το συνέδριο. Νομίζω ότι πραγματικά είναι πραγματικά πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε την εφαρμογή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη συμμετοχή και ευρωβουλευτών αλλά και των εθνικών βουλευτών για όλους τους λόγους που ανέφεραν οι προηγούμενοι μιλητές. Είμαι πρόεδρο τη ε, ομάδα εργασία του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά ανθρώπινα δικαιώματα σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο παρελθόν ε, Έχω εμπειρία σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, σε ό,τι αφορά και τη συμμετοχή μου σε Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων των Εθνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βέβαιος ότι και οι διαστάσει είναι πάρα πολύ σημαντικέ σε ό,τι αφορά την κατάρτιση μια αποτελεσματική πολιτική ή τα ανθρώπινα δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ασφαλώ για τα ανθρώπινα δικαιώματα τη Λισαβόνα τον είσαι Και θα πρέπει η συνθήκη της Λισαβόνας τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο τη εργασια μα. Μου ζητήθηκε να επικεντρωθώ στο έργο μου στα πολυμερή φόρα, κυρίως τον ΟΙΕ. Θα το κάνω αυτό, θα καλύψω τρία σημεία, θα πω λίγο παραπάνω ε, λόγια αν θέλετε για τους ελέγχους της ΚΟΓΟΜ, να σας εξηγήσω πώς προσπαθούμε να ε, βελτιώσουμε το έργο μας και από πλευρά μου θα ήθελα να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις για, για το ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων σε ό,τι αφορά το ρόλο της ΚΟΧΟΜ. νόματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε το 1987 για να βελτιωθεί ο συντονισμός κατά βάση μεταξύ των, μεταξύ των ε, κρατών μελών. Το του Συμβουλίου Εκτορικών Υποθέσεων να προετοιμάσει λοιπόν ε, τις αποφάσεις του ε, Συμβουλίου είναι σκοπός μας και ασφαλώς μεταβιβάσει τέτοια μηνύματα. Μία σημαντική αλλαγή ε, σε ό,τι αφορά την εργασία του Συμβουλίου και τον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων και τα ανθρώπινων δικαιώματα σημειώθηκε κατά την ε, υπογραφή της συνθήκης της Λισαβόνας. Έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Άρα τώρα οι υπάλληλοι Τη εξωτερική υπηρεσία δράση τη Υπηρεσία εξωτερική δράση προεδρεύουν των ομάδων εργασίας μας. Άρα αντικαταστάθηκε η εξαμηνία εκπεριτροπή προεδρία πλέον από την Υπηρεσία εξωτερική δράση. Δεν... Τώρα λοιπόν είναι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αυτή που καθοδογεί τις εργασίες του Συμβούλιο και σε αυτή την κατάσταση είναι ακόμα πιο σημαντική η προσωπική δέσμευση των κρατών μελών. Επίσης αυξήθηκε το φορτίο εργασίας με την πάροδο των χρόνων. Αρχικά συναντιόμαστε μόνο δύο φορές κάθε χρόνο για να προετοιμάσουμε το έργο μας. Τώρα συναντιόμαστε τακτικά και με εκπροσώπους από τις πρωτεύουσε, αλλά όπως σας είπα και με τους υπαλλήλους που εδρεύουν στις Βρυξέλλες. Υπάρχει μία μόνιμη επιτροπή στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ στις Βρυξέλλες. Αυτό ήταν μία απόρρια του στρατηγικού πλαισίου. Πέρσι συναντηθήκαμε στη Γενέβη στις αρχές του έτους με τους πρέσβεις και τους εκπροσώπους των κρατών μελών για να προετοιμάσουμε το έργο μας σε επίπεδο ΟΗΕ. Η Κόχομ λοιπόν αντιμετωπίζει το πλήρες φάσμα των θεμάτων ανθρωπινών δικαιωμάτων και εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήρες φάσμα. Αλλά περιορίζεται στην εξωτερική δράση. Δεν έχει επίσημη εντολή να συζητά θέματα εσωτερικά στο Κοινοβούλιο. Είναι κάπως παρόμοιο με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και εξωτερικών υποθέσεων στο Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια αντιστοιχία. Όπως είπε και ο Σταύρος προηγουμένως, υπάρχει το θέμα της εσωτερικής και εξωτερικής συνέπειας και συνοχής στην δράση μας και αυτό ως θέμα είναι όλο και πιο κρίσιμο για την αξιοπιστία μας και την εγκυρότητα μας και σε διμερές αλλά και σε πολυμερές επίπεδο. Αυτό λοιπόν πραγματικά μας απασχολεί όλο και πιο πολύ. Να πω ότι κάποια από το έργο μας τα τελευταία χρόνια ήταν η διαπραγμάτευση του θεγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης και η σχετική εντολή εγκρίθηκε πέρσι, αλλά και σχετικές ε, κατευθυντήριες γραμμές. Όπως αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην κατάσταση αυτή, ο ρόλος των κρατών μελών παραμένει κρίσιμος. Όχι ε, μόνο επί τα θέματα που αφορούν την ε, ασφάλεια και τις εξωτερικές υποθέσεις χρειάζονται ομοφωνία, αλλά γιατί θέλουμε πλήρη δέσμευση και διακτησία από πλευρά των κρατών μελών θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πλήρη συνδέσμευση για την εφαρμογή της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και από πλευρά ικανοτήτων σε ό,τι αφορά την κατανομή των ευθυνών. Υπάρχουν ε, έντρες όπως η Γενέβη, η Ζηρίχη, το Στρασβούργο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΟΗΕ, εδώ, όπως ε, αναφέρεται και στο στρατηγικό πλαίσιο άλλωστε, το οποίο εγκρίθηκε πέρσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη σημασία σε ένα λειτουργικό σύστημα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να υπάρχουν υψηλά πρότυπα παγκοσμίω, ναι. αλλά και μηχανισμοί που διασφαλίζουν την εποπτεία τη εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ σκληρά εργαστήκαμε προκειμένου το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να καταστεί ένα αξιόπιστο σώμα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης. Η βασική στόχη είναι η ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα του ΥΠΑ του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποστηρίζεται και οικονομικά με σημαντικό τρόπο η καθολικότητα της ε, περιοδικής αναθεώρησης και το καθεξής. Επίσης, προκειμένου να είναι καλύτερη η δουλειά μας, στα φόρα του ΟΗΕ, ιδιαίτερα στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ξεκινάμε μια στρατηγική συζήτηση και προετοιμασία των διαφόρων συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από πέρσι λοιπόν προετοιμάζουμε τις συνεδριάσεις για όλες τις τακτικές μάλλον συνεδριάσεις της Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το σημείο κίνησης είναι πάντα η κοινή συνάντηση της ΚΟΧΟΜ και των ε, πρέσβεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην Γενέβη. Άρα εκεί εντοπίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ποια είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία ε, καταγράφονται σε ένα έγγραφο στρατηγικής εσωτερικό και δημοσιεύονται και σχετικά ε, συμπεράσματα του Συμβουλίου το Φεβρουάριο. Και αυτό ασφαλώς επηρεάζει το έργο μας και πάντα φυσικά υπάρχουν και θέματα που ανακύπτουν τελευταία στιγμή έκτακτα γεγονότα. Έχουμε λοιπόν πάντα δύο-τρει προτεραιότητε, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε πάρα πολλέ προτεραιότητε και να χανόμαστε. Εντοπίζουμε κάποιε προτεραιότητε, κάποιε πρωτοβουλίε, ε, κοιτάμε τι πρωτοβουλίε υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο, προετοιμαζόμαστε καλύτερα για θέματα για τα οποία βρισκόμαστε σε αμυντική στάση και είμαστε έτσι σε καλύτερη θέση να προετοιμάσουμε τη συνέδριση και έτσι μπορούμε να επιδιώξουμε μια σειρά προτεραιοτήτων στον ΟΗΕ. Τώρα, στην παρούσα φάση έχουμε χώρες όπως ε, η Συρία, η Λευκορωσία, η Βερμανία, η Μιανμάρ, η μεταβατική αυτή φάση, αλλά και θεματικά θέματα όπως η θαντική καταδίκη και τα δικαιώματα του παιδιού, η ελευθερία έκφρασης και το καθεξής. Επίσης, σε ό,τι αφορά το καθεστώς των γυναικών, υπάρχει το σχετικό σώμα του ΟΙΕ για την ενίσχυση του κεκτημένου σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και τις ισότητες των φύλων. Και βλέπουμε ότι μέσω του έργου μας είμαστε σε καλύτερη θέση να ξεκινήσουμε εγκαίρως ε, συνεργασία με τρίτα κρατημέλη Όπω καταφέραμε για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την θανατική καταδίκη, πλέον είναι ένα θέμα το οποίο έχει καθιερωθεί σε επίπεδο ΟΗΕ και λαμβάνουμε την υποστηρίξη του ΟΗΕ. Επίσης, ε, με το στρατογικό προγραμματισμό καταφέρουμε να βάζουμε θέματα στην ατζέντα, όπως για παράδειγμα το θέμα της Λευκορωσίας. Αλλά και να προετοιμάσουμε καλύτερα τι θέσει μα για θέματα όπου δεν είχαμε τοποθέτηση ε, στο παρελθόν, ήταν διστάμενες οι απόψεις, όπως για παράδειγμα οι ιδιωτικέ ε, εταιρείε για την ε, αποστολή στρατιωτών. Και σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη διαχείριση των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνεκτική, γραπτή έκθεση. Θα ήθελα επίσης... Ναι, ναι, βλέπω το ρολόι. Έχω 20 δευτερόλεπτα. Έχω μόναχα λίγα σημεία τα οποία θα σας αναφέρω από τη δική μου εμπειρία. Κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τη συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μερικά θέματα που έχουν να κάνουν με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όπως ανελέχθη ήδη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως στο πολυμερές πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις σχέσεις με τον ΟΗΕ. Η Πατή εκπρόσωπος προσπαθεί να αντιμετωπίζει πάντα τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην, ε, στα πλαίσια του ΟΗΕ το κάνουν και άλλες μεγάλες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ. και όπως ανέφερα και στην ΚΟΧΟΜ η ομάδα εργασίας αυτής είναι το μόνο, η μόνη εργασία του Συμβουλίου που μετά από κάθε συνάντηση έρχεται σε επαφή και με ΜΚΟ και με εκπροσώπους Συμβουλίου της Ευρώπης και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να τους κρατήσει ενημέρωση για τις εξελίξεις. Για μας ο λόγος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ψήφισμα που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε χρόνο σε σχέση με τις προτεραιότητες για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα σημαντικό έγγραφο αναφοράς. Το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά αυτές τις πρωτοβουλίες και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Ολομέλεια είναι μια σημαντική συμβολή στη διατύπωση πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίσκεψη κάθε χρόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενέβη είναι ένα σημαντικό θέμα. Με τον τρόπο αυτό οι χώρες της, ε, του ΟΗΕ μπορούν να έχουν μια σαφή ιδέα για τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το ενδιαφέρον που δείχνει για τα τεκτενόμενα και φυσικά είναι σημαντικές οι θέσεις που εγκρίνει. Έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις σημαντική υποστήριξη από το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο παραγωγός σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες να υπάρξει πρόοδος όπως το, τα δικαιώματα των ε, ΛΙΑΔ. ΛΟΑΤ, Το γεγονό ότι τα θέματα αυτά τίθενται και σε συναντήσει μεταξύ τη αντιπρόσωπη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου τη Νότια Αφρική και αυτό ήταν μια πολύ σημαντική συμβολή στη συζήτηση. Ένα τελευταίο σημείο, ένα σημαντικό στοιχείο για να χρησιμοποιηθεί να χρησιμοποιηθούν τα πορίσματα του Μηχανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να τους δώσει κανείς ορατότητα και πολιτική εμβέλεια. Αυτό γίνεται με τις ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ειδικού εισηγητές από το Ηνωμένα Έθνη και άλλους φορείς. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ λοιπόν και εμείς να έχουμε επαφή με αυτούς τους μηχανισμούς. Θα μας ενδιαφέρει επίσης να ακούσουμε και την άποψη των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων αν έχουν αντίστοιχε εμπειρίες για τους μηχανισμούς που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γέννη και τη συνεργασία με πολυμερή φόρα. Από την δική πλευρά, όπως είπα και προηγουμένω είναι κέρδιας σημασίας οποιαδήποτε συζήτηση που γίνεται σε εθνικό επίπεδο για την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων να διατηρεί σαν σημαντικό ε, στοιχείο την εφαρμογή της πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τόνισε το στρατηγικό πλαίσιο, τόνισε την κοινή ευθύνη της Ευρωπαϊκής και των κρατών μελών και έχει αποφασίσει ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο και τα κράτη-μέλη μεμονωμένα μπορούν στεναρά να εγείρουν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους διμερείς διαλόγους και στο ύπατο επίπεδο επίσης. Προφανώ προφανώς δεν γίνεται αυτό πάντα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε μια μεγαλύτερη πρόοδο στα θέματα αυτά. Το στρατηγικό πλαίσιο επίση περιλαμβάνει μια δέσμευση των κρατών μελών να δώσουν το καλό παράδειγμα με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο, στο εσωτερικό τους. Πάντα τίθεται το ερώτημα πώς εμείς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι παρακολουθούμε πλήρως τα συμπεράσματα και εφαρμόζουμε τις απόψεις των ειδικών εισηγητών και αντιμετωπίζουμε όλες τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν πολλά θέματα λοιπόν τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας και σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τόιερμαν για τη λεπτομερή σας παρέμβαση. Στρέφουμε προς εσάς, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που έθεσε ο κύριος Στόιερμαν και είναι πολύ ενδιαφέρον ε, να ακούσουμε και από εσά, ε, από τα Εθνικά Κοινοβούλια, αν και κατά πόσο παρακολουθείτε μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών σας ε, τι ακριβώς γίνεται στην ομάδα Κοχόμ, είτε και απευθείας στη Γενέβη ή στη Νέα Υόρκη. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Υποθέτω κύριε Τόιερμαν ότι όταν ήμασταν στη Γενέβη μου έκανε εντύπωση ότι άκουσα από, από πολλούς διπλωμάτες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το ότι χαιρετίζουν ε, το γεγονός ότι οι διπλωμάτες έρχονται σε ένα τέτοιο πολιτικό φόρουμ για να ε, υποστηρίξουν αυτό που κάνουν ε, οι ε, διπλωμάτες σε εθνικό επίπεδο. Είναι γεγονός ότι είναι μερικά ζητήματα που είναι δύσκολο να τα διαχειριστεί κανείς, πάντως είναι ευπρόσδεκτη. Οπότε θα ήθελα, αν σε εθνικό επίπεδο εργάζεστε επί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να πάτε σε τέτοιου είδους φόρα, ακόμη και αν είναι μακριά, ε, γιατί συζητούν ψηφίσματα τα οποία δεν τα μαθαίνει κανείς σε εθνικό επίπεδο ή ε, πολιτικώς αμφισβητούμενα ψηφίσματα. Ε, σας ενθαρρύνω λοιπόν να μεταβείτε. Στην αρχή στις Βρυξέλλες εδώ είχαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ υποστήριξη από, το, ε, από την ομάδα του ΙΠΑ του Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, όταν αρχίσαμε τη δουλειά μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα μας βοήθησαν πολύ να διαμορφώσουμε την πολιτική μας και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρσι αποφάσισε να χρηματοδοτήσει περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί ε, τους φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί όλο και περισσότερο διευρύνεται το φάσμα της εργασίας τους, έχουν όλο και περισσότερα γραφεία στις διάφορες χώρες και έχουν όλο και περισσότερα πράγματα να κάνουν και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα έπρεπε οποιοδήποτε συμμετέχει σε αυτή τη δουλειά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να τους ε, συνεπικουρεί θα έπρεπε να ε, εστιάσουμε την, ε, τις εργασίες μας σε μια πιο οικουμενική προσέγγιση. Δεν θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Yes, uh, actually I I give you the floor, but can't see. Να σας δώσω το λόγο, αλλά δεν βλέπω το όνομά σας. Μήπως μπορείτε να μας πείτε, να μας συστηθείτε. Jina Marlin Farrugia mill-Parlament tar-Repubblika ta' Malta. Waqt li η κυρία Φαρούτζα από το ε, Κοινοβούλιο της Μάλτας. Συμφωνούμε όλοι ότι όταν ένας άνθρωπος γεννιέται, γεννιέται ε, στην αξιοπρέπεια, με ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και με υποχρεώσεις και ευθύνες Τα ανθρώπινα δικαιώματα όμως μπορεί να παραμείνουν θεωρία αν δεν τα ε, υλοποιούμε. Άκουσα τις διάφορες ομιλίες, ε, έχω διαβάσει πολύ, όλοι σας θα έχετε παρακολουθήσει το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πρόβλημα της έλλειψης σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους ε, διάφορους φορείς, ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, υπόθηκε και αυτό, πρέπει να ενισχυθούν, η, η κοινωνία των πολιτών επίσης, για να μπορέσει όμως ένας άνθρωπος να γνωρίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, τους, πρέπει, τις υποχρεώσεις του, πρέπει και εμείς να αρχίσουμε με μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση και γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τις εκπαιδευτικές υποδομές, ε, ε, τα σχολικά προγράμματα ε, σε εθνικό επίπεδο. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, ώστε εξαπαλώνων ήχων τα παιδιά να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους που δεν πρέπει να παραμείνουν νεκρό γράμμα, πρέπει να είναι γνωστά. Να ξέρει ο κάθε άνθρωπος ποια είναι ε, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του. Αυτό πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα της ύπαρξής του. Επειδή πρέπει να συνεχίσουμε να... Ε, ε, να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα προβλήματα, ε, πρέπει, να απαραίτητη πρόληψη για τις επόμενες, ε, τις μελλοντικές γενναίες. πρέπει να διαμορφώσουμε αυτούς τους νέους ηγέτες ε, από την, από, από την παιδική τους ηλικία ήδη να γνωρίζουν αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για να μπορέσουμε να ε, μπούμε στην ουσία του προβλήματος. Ευχαριστούμε όλους όσους ε, έλαβαν το λόγο και όλους τους προσκεκλημένους για τις παρουσιάσεις, γιατί μας βοηθούν να δούμε το πρόβλημα πιο ε, πολύπλευρα. Πρέπει να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα όχι βραχυπρόθεσμα, γιατί οι μελλοντικέ γενναίες θα προκύψουν από τα σημερινά παιδιά και πρέπει να τα μορφώσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε ο κόσμος να είναι καλύτερος για όλους. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την έκκληση που κάνατε επίσης να υπάρξει μια κουλτούρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την παιδεία σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχω τα στοιχεία στα χέρια μου, ξέρω ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται στις εξωτερικές σχέσεις για παιδεία στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημιουργία ενός κλίματος και μιας κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μου επιτρέπετε. Να συνεχίσω αυτά που είπατε. Νομίζω ότι κάθε άτομα έχει ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και καθήκοντα που έλκονται από αυτά. Όλοι ως πολίτες έχουμε το καθήκον <clears throat> να σεβόμαστε τον νόμο. Αλλά υπήρξε πριν από κάποιο διάστημα μια συζήτηση και αυτό είναι ένα ερώτημα προς τον κύριο Τόιερμαν. Μια συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιωμάτα και πολλές χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαν μέσα στα πλαίσια της φιλοσοφικής αυτής συζήτησης ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να παρέχονται μονάχα στα άτομα τα οποία τηρούν τα καθήκοντα που προέρχονται από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι κάτι το πολύ υπερβολικό. Έχει κάνει ανθρώπινα δικαιώματα ως ανθρώπινο ακόμα και αν είναι εγκληματίας. Και θυμάμαι ότι στο παρελθόν υπήρχε μια προσπάθεια να αφαιρεθεί το θέμα αυτό από, τα, από την ατζέντα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα ήθελα να ξέρω και από εσά λοιπόν κύριε Τόεμαν αυτή είναι μια συζήτηση που θα επανέλθει ή έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Για το ερώτημα που αναφέρατε για την εκπαίδευση σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις άλλες δραστηριότητε, δεν είναι... Μπορώ να σας δώσω αριθμητικά στοιχεία, αλλά νομίζω ότι και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι θα ήταν πιο ειδήμονες στο θέμα αυτό. Να πω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Πλαισίου και του Σχεδίου Δράση. Προσπαθούμε να συνενώσουμε το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων προκειμένου να έχουμε πολλά εργαλεία στη διάθεσή μα, Γιατί ουσιαστικά το πιο μεγάλο έργο θα πρέπει να συμβεί σε επίπεδο κράτους εθνικού. Και θα πρέπει να υποστηριχθεί η τοπική κοινωνία των πολιτών να υποστηρίξει με τη σειρά της το έργο των κυβερνήσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συμβάλλουμε και σε μια κουλτούρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η υποστήριξη στον τομέα της παιδείας, αλλά να συμπεριληφθούν και θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων στην παιδεία. Κρίσιμη σημασία είναι αυτό σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, υποτροφίες, κάποια μάστερ τοπικά. Να σας πω ότι εγώ τότε είχα σπουδάσει στην Ευρώπη, αλλά και τότε που σπούδασα εγώ ήταν πάρα πολύ λίγα τα προγράμματα που ήταν αφιερωμένα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχουν πολλές δραστηριότητε σε πολλές περιφέρειες που πραγματικά όλα αυτά θα ενδυναμώσουν την κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό που αναφέρατε είναι η συζήτηση για τα δικαιώματα και τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις. Αυτή η συζήτηση όντω έχει ανακύψει σε διάφορες περιστάσεις κατά το παρελθόν. Δεν είναι συζήτηση που κάνουμε στην παρούσα φάση το θέμα που αναφέρθηκε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την 50η επέτειο της συνθήκη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε ό,τι αφορά και τα, τις σχετικές υποχρεώσεις, δεν ε, συνεχίστηκε το θέμα αυτό. Αλλά η όλη συζήτηση ε, εντάσσεται σε μια πιο ευρεία πρόκληση. Το όλο θέμα της ε, διατήρησης της καθολικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλές δραστηριότητες υπάρχουν και τα τελευταία 10-15 χρόνια. Αν συγκρίσουμε πόσες επικυρώσεις ε, γίνονται σε ό,τι αφορά μεγάλες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι πραγματικά εντυπωσιακή η πρόοδος. Αλλά εξακολουθούμε να βλέπουμε το εξής, ότι πολλές χώρες εξακολουθούν να έχουν πάρα πολύ μεγάλες επιφυλάξεις, επίσης πολιτικά επιχειρήματα και προκλήσεις σε ό,τι αφορά την καθολικότητα. Εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ στεναροί. Ένα βασικό στοιχείο σε όλα αυτά είναι ότι οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ή ως Ευρωπαϊκές χώρες είναι όχι μόνο να διαπραγματευόμαστε με χώρες ε, για τα θέματα αυτά, αλλά να ζητούμε και την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την βιώσιμη διαμόρφωση της καθολικότητας. Επιτρέψτε μου να κάνω και μία προσθήκη σε ό,τι αφορά και τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να σας πω ότι το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία περιλαμβάνει μία σειρά σημαντικών δεσμεύσεων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη με σκοπό να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ηγετική σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των ε, κατευθυντηρίων γραμμών, για παράδειγμα, για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρθηκε. Αναφέρθηκαν τα σχετικά βήματα που έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κατεύθυνση αυτή σε ό,τι αφορά τη δέσμευση ανάληψη σημαντική δράση προκειμένου όλα αυτά να ενταχθούν στις πολιτικές μας, αλλά είναι σημαντικό επίσης ότι στο σχέδιο δράσης όλα τα κρατημέλη δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν και ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τις επιχειρήσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι, ερμηνεύοντας και μεταφέροντας σε εθνικά σχέδια δράσης αυτές τις ε, κατευθυντήριες γραμμές για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. σκοπός μας είναι να το έχουμε πετύχει αυτό μέχρι το τέλος του έτους. Μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά κάποια κρατημέλη το έχουν ήδη πράξει αυτό. Σε κάποια άλλα συνεχίζεται η δουλειά. Είναι σημαντικό ο τομέα αυτό σε κάθε περίπτωση για την ενεργό συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιατί όντω, όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι τη δουλειά μα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιο άλλο που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ίσως υποθέτω ότι η σιωπή σας δεν είναι και η απάντηση για το αν απαντάτε στο ερώτημα στα εθνικά σας κοινοβούλια, στο ερώτημα των πολιτικών που ακολουθούν οι κυβερνήσεις σας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Γενέβη. Δεν κάνετε, δεν ασχολείστε λοιπόν με το θέμα αυτό. Εάν δεν το πράτετε θα σας παροτρύνω να το πράξετε στο μέλλον. Να σας δώσω ένα παράδειγμα ακόμα. Στην προηγούμενη ε, συζήτησή μας είχαμε ακούσει από τις κοινωνίες των πολιτών πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε τις ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μεγάλες χώρες όπως η Ρωσία ή η Κίνα, όπου υπάρχουν και άλλα οικονομικά συμφέροντα τα οποία εμπλέκονται. Η περίπτωση Μαγνίτσκη, όπου φυλακίστηκαν και οι συνήγοροι του κατηγορουμένου υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν από πού προέρχονται όλες αυτές οι ενέργειες και ποιος είναι υπεύθυνο για όλα αυτά. Θα μπορούσε να υπάρχει μια απόφαση από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουμε συνέχεια σε αυτήν την περίπτωση και να πούμε ότι τα άτομα αυτά <clears throat> για την δολοφονία του κρατουμένου, για τον θάνατο του κρατουμένου στη φυλακή του Μαγνήσικη, θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε κυρώσεις εναντίον των ατόμων αυτών και να ε, παγώσουν τα στοιχεία ενεργητικού τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. σε σχέση με τα θέματα αυτά υπήρξε μόνο μία απάντηση από ένα κράτος μέλος για το τι πιστεύουν για το θέμα αυτό. Υποθέτω ότι αν οι διπλωμάτες αυτοί ακούγαν από εσάς τους ε, εκλεγμένους βουλευτές στις χώρες τους, και ξέρω ότι πολλές χώρες παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή την κατάσταση στη Ρωσία και οι εκλεγμένοι βουλευτές και η κοινή γνώμη, τότε θα μπορούσε ίσως να προκύψει μια μεγαλύτερη πίεση προς τους διπλωμάτες στην ΚΟΧΟΜ να έχουν μια πιο στεναρή Δεν βλέπω το όνομά σας όμως. Αν θέλετε να παρουσιάσετε τον εαυτό σας, σας δίνω τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε και κάποιο κίνητρο για να λάβω το λόγο. Η, το Ιταλικό Κοινοβούλιο έχει ιδιαίτερη δέσμευση για τα θέματα αυτά που συζητούμε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε πρόκειται για τον χώρο εκτός, εξωτερική, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε για το εσωτερικό μέτωπο. Έχουμε μια Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Βουλή των Αντιποσώπων και στη Γερουσία και συμμετέχει ιδιαίτερα στα τεκτενόμενα των ε, ευρωπαϊκών θεσμών εγώ είμαι μέλος της αντιπροσωπείας της Ιταλίας στο Συμβουλίο της Ευρώπης όπου συζητάμε πολλές περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία με μεγάλη δέσμευση της χώρας μας στα διεθνή φόρα για τα θέματα αυτά και στο Κοχόμ στη Γενέβη ιδιαίτερα στην τρέχουσα θητεία η οποία ξεκίνησε την άνοιξη του 2013 το νέο μας κοινοβούλιο έχει αποδώσει μια ιδιαίτερη προσοχή που έχει εκφραστεί πολλές φορές και από την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της κυρίας Μπολτρίνη σε δημόσιες ε, δηλώσεις δίνουμε ιδιαίτερη σημασία να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ της εξωτερικής μας πολιτικής και της εσωτερικής μας πολιτικής γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ελεγχτούμε η Ευρώπη η οποία έχει αποτελέσει το λίκνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αγωνίζεται για να μπορέσουν να προσπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες, ότι αυτή η ίδια Ευρώπη δεν σέβεται αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της. Γι' αυτό το, Ευρωπαϊκό μας, <clears throat> το Εθνικό μας Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει μια σειρά από ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης στο εσωτερικό της χώρας μας για την εφαρμογή της νομοθεσίας και αναφέρομαι περισσότερο στην συζήτηση που προέκυψε για τους κρατούμενους στα σοφρονιστικά ιδρύματα, την περίπτωση των ατόμων ΛΟΑΔ και έχουμε σε συζήτηση ένα νόμο κατά της ομοφοβίας και της φοβίας των μεταφυλικών ατόμων, επίσης η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Τόιρε στην ε, παρέμβασή του, το θέμα της αντιμετώπισης των μεταναστών και η σύνδεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σύνορά της και σε σχέση με αυτό το θέμα περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια πιο ομοιόμορφη μεταχείριση. Είναι ένα κλασικό θέμα όπου είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε τη συνεκτικότητα όλων αυτών των ενεργειών και την αλληλεγγύη και υποστήριξη προς τις χώρες οι οποίες έχουν σύνορα πιο εκτεθειμένα στα μεταναστευτικά φαινόμενα. Κάτι ακόμα που θέλω να υπογραμμίσω. Βλέπω ότι υπάρχει σημαντική έμφαση που δίνεται στο θέμα αυτό της συνεκτικότητος, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο να είμαστε αξιόπιστοι από ότι να αντιμετωπίσουμε τις συγκεκριμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει με να είμαστε αξιόπιστοι, αλλά πιο πολύ προέχει το να προστατεύσουμε τη ζωή των ατόμων και τα ψηφίσματά μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει πολύ συχνά μια έμφαση στην υποστήριξη των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ νομίζω ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι εξίσου ή υπέρτερη σε σημασία με την προάσπιση των αξιών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πηγάζουν από τις συγκεκριμένες εμπειρίες και τα βάσανα πραγματικών ανθρωπίνων όντων και δεν είναι μοναχαφηρημένα. Ένα δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε και ίσως το απόγευμα θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό για τις ενδεχόμενες κυρώσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εφαρμόσει όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό της. Μου φαίνεται λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε <clears throat> πώς το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται στο εσωτερικό μιας κοινωνίας των πολιτών που μπορεί να αναγνωρίσει και να γίνεται αναγνωρίσιμη ως, αντικείμενο ως υποκείμενο δικαίου, ως νομικό και ηθικό πρόσωπο. Θέλω λοιπόν να εξασφαλίσω ότι αυτή η δράση της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να συμπληρώσει ή να παίξει σημαντικό ρόλο πέραν των σχέσεων πέραν των κυρώσεων. Επομένως θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο τις οριζόντιες συνδέσεις και όχι μοναχά τις κάθετες επιβολές. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Κύριος Νικολέτη. Και έχω δύο συναδέλφους που λέγονται, ευχαριστώ τον κύριο ε, Νικολέτη, και έχω δύο ομιλητέ με το όνομα Γκόμε, τον κύριο Γκόμε από το Ισπανικό Κοινοβούλιο και μετά την κυρία Γκόμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα την Πορτογαλία. Ο κύριο Γκόμες. Σας ευχαριστώ. Θέλω να σας εκθέσω δύο σκέψει. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με τη δράση των κυβερνήσεων των κρατών μελών όταν πρόκειται για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ισπανική κυβέρνηση το 2008 ενέκρινε ένα εθνικό σχέδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο τέλος του 2013 θα παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο εθνικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα με στόχο να αναζωογονήσει, να συμπληρώσει το θεσμικό και συνταγματικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ισπανία. Αυτή η ενημέρωση του εθνικού σχεδίου έχει σαν στόχο όλες οι αποφάσεις σε επίπεδο κοινοβουλευτικό ή σε επίπεδο κυβερνητικό να διατρέχονται από το πνεύμα αυτού του εθνικού σχεδίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρθηκε η περίπτωση Μαγνίσκη και η περίπτωση του Ρώσου συνηγόρου ο οποίος ε, βασανίστηκε και στο τέλος έχασε τη ζωή του σε μια φυλακή της Ρωσίας. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχόλησε πολλούς ε, διεθνείς φορείς όπως και τον ΟΑΣΕ στον οποίο εγώ συμμετέσχα σε μία ε, συνάντηση αλλά υπήρξαν και πολλά κάποια κοινοβούλια αυτή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν πιο ευαίσθητα από άλλα σε αυτή την πολύ συγκεκριμένη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξε ιδιαίτερη ενεργητικότητα για το θέμα αυτό. Στην Ευρώπη ήταν το Αγγλικό Κοινοβούλιο, το Βρετανικό Κοινοβούλιο και το Ισπανικό που υποδεχτήκαμε ένα εκπρόσωπο του κ. Μαγνίσκη και είχαμε μια συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Θεμάτων. Αλλά έπαιξαν άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, εθνικά κοινοβούλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δεν ήταν τόσο ευαίσθητα στο θέμα αυτό και δεν προέβησαν σε κάποια συζήτηση για τα θέματα αυτά. Γι' αυτό θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στην ανάγκη να υπάρχει μια μεγαλύτερη αλληλεγγύη και συνοχή μεταξύ των, Ευρω... των κοινοβουλίων της Ευρώπης όταν αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα. Γιατί πολλές φορές εμπλέκονται οι οικονομικά συμφέροντα τα οποία εμποδίζουν την καταγγελία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και επειδή υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πνεύμα στις παγκόσμιες αγορές, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα ενιαίο πρότυπο προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα έπρεπε τα θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουν μια μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Το δεύτερο θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι κάτι το οποίο ήδη έχει φύγει <clears throat> στις προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε σήμερα το πρωί και εδώ αναφέρομαι στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα κράτη-μέλη μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένες παραβιάσεις που μπορούν να γίνουν λόγω κατάχρησης εξουσίας, λόγω παράνομε, παράνομων ενεργειών, αλλά αναφέρομαι τις διαρθρωμένες μορφές παραβιάσεων που μπορούν να λάβουν χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και είναι μια από τις θεμελιώδες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο πολιτικός ε, πλουραλισμός είναι μια βασική εγγύηση <clears throat> για τη δημοκρατία. Και από την απαρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πριν, υπήρχαν πάντα οι εχθροί της ανοιχτή κοινωνίας, για να χρησιμοποιήσω τη φράση του Πόπερ, αυτοί οι εχθροί της ανοιχτή κοινωνίας και της δημοκρατίας ήταν πάντα από τη μια μεριά ο ολοκληρωτισμός και από την άλλη πλευρά η κινήσεις οι οποίες βασίζονται σε μια ριζοσπαστική αναζήτηση ταυτότητας. Μη δημοκρατικά λοιπόν κινήματα που διεκδικούν μια ταυτότητα. <clears throat> Πρέπει λοιπόν μέσα στο σχέδιο δράσης να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς τους αντιπάλους της ανοιχτής κοινωνίας. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση όταν και λόγω της οικονομικής κρίσης και των κοινωνικών επιπτώσεων ε, υπάρχει η αναζωπήρωση ορισμένων πολιτικών σχηματισμών που είναι σαφώς εξτρεμιστικοί σε σχέση με την εθνική ταυτότητα ή ολοκληρωτικοί και έχουν σαν στόχο να ε, υπονομεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. <clears throat> Μιλήσαμε για την κοινωνία των πολιτών, αλλά όπως ελέγχθηκε σε μια προηγούμενη ε, παρέμβαση υπάρχει η κοινωνία των πολιτών που έχει αυθόρμητο χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν και οργανισμοί στην κοινωνία των πολιτών που εξυπηρετούν τους σκοπούς κομμάτων τα οποία είναι αντιδημοκρατικά. Θα με ενδιαφέρει να υπάρχει μια περισσότερη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Η Άννα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Ραμόν Χουαρεγκέ ανέφερε και στη δική του παρέμβαση σε ό,τι αφορά τη σημασία που έχει το να εξεταστεί ο ρόλο των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την προώθηση ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου ότι όλε οι πτυχέ που αφορούν την εταιρική ε, ευθύνη, κοινωνική ευθύνη να εξεταστούν. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για το έργο μα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό ρόλο για τα εθνικά κοινοβούλια να υπενθυμίσω τη σημασία της ε, σύμβασης κατά της διαφθοράς. Να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να περάσει εθνική νομοθεσία για να αντιμετωπιστούν τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Νομίζω ότι βλέπουμε να αναδύεται ένα νέο επίπεδο σύνδεσης σαφούς μεταξύ της διεύρυνσης και της ε, διαφθοράς και της παραβίασης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να καλυφθούν, να συγκαλυφθούν αυτές ε, οι περιστάσεις, οι υποθέσεις διαφθοράς. Αυτό το έχουμε δει σε διάφορες περιστάσεις, για παράδειγμα στην Αγκόλα. οι πιο πολλές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων και των επιθέσεων κατά των ακτιβιστών και των δημοσιογράφων σχετίζονται άμεσα με την απόπειρα να τους φημώσουν για να μην καταγγείλουν περιστατικά διαφθοράς και σημαντικές διαφθορές, συγγνώμη, παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και με την παγκοσμιοποίηση, με την κρίση στον κόσμο, βλέπουμε τυχοδιώκτες και εκατομμυριούχους στην Αγγόλα να αγοράζουν, για παράδειγμα, στην Πορτογαλία τον τύπο. Όχι μόνο για το κύρος που τους δίνει αυτό, αλλά για να φημώσουν τα μέσα ενημέρωση στην Ευρώπη, στην Πορτογαλία, για αυτά που συμβαίνουν για τις παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Αγγόλα και βλέπω ότι μιλώντας με τους Πορτογάλους δημοσιογράφους που εκφοβίζονται λόγω της κρίσης φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. Και το βλέπω μπροστά στα μάτια μου να συμβαίνει. Δεν ε, προβαίνουν σε τέτοιες ε, καταγγελίες και αυτό είναι χειρότερο από όλα. Το χειρότερο από όλα αυτή η αυτολογοκρισία και αυτό που είπε η κυρία Λοχμπίλερ είναι πολύ σημαντικό ότι εδώ τώρα στο Κοινοβούλιο μιλάμε για θέματα διαφθορά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει περάσει αυτό από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα πάει στην Ολομέλη την επόμενη, στην επόμενη σύνοδο. Και καλό λοιπόν τα Εθνικά Κοινοβούλια να δουν τι μπορούν να κάνουν σε εθνικό επίπεδο για να εφαρμόσουν τις πτυχές αυτές. Να πω επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της ΚΟΧΟΜ. Η ΚΟΧΟΜ και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η Αντιπρόεδρος και ο ύπατος αρμοστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει όλοι αυτοί να συντονιστούν πολύ καλύτερα και θα πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμό των τομεακών πολιτικών, να υπάρχει μια ενιαία πολιτική που θα συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά αυτό το φροντίζει ο Σταύρος Λαμπρινίδης αλλά χρειάζεται πολιτική καθοδήγηση σε πολύ υψηλό επίπεδο και δεν βλέπουν να, το, να γίνεται κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, υπάρχουν τρία, τρεις ε, υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυλακισμένοι στο Μπαχρέιν. Το είπε αυτό η Human Rights Watch. Οι ευρωπαϊκές αρχές κάνουν εκστρατείες για τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ξεχνούν τέτοιους ε, υπηκόους που είναι στη φυλακή, για την Αιθιοπία για παράδειγμα. Κινητοποιηθήκαμε για να βγάλουμε δύο Σουηδούς δημοσιογράφους. Αλλά τι κάναμε για τους χιλιάδες δημοσιογράφους και τους ακτεβιστές που είναι φυλακισμένοι στην Αιθιοπία και μιλάμε για μια χώρα πάρα πολύ σημαντική στην Αφρική. εταίρο μας στην κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση με τις χώρες ΑΚΕ. Μια χώρα όπου πραγματικά έχουμε επιρροή. Και πολύ απλά δεν κάνουμε τίποτε. Θα πρέπει λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα να ενταχθούν στις πολιτικές μας, στις εμπορικές μας πολιτικές, στις αναπτυξιακές μας πολιτικές και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δύο τελευταία θέματα θα ήθελα να αναφέρω και θα πρέπει να συνεργαστούμε από αυτόν με τους συναδέλφους μας σε ό,τι αφορά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Βλέποντας ε, τις εκστρατείες των εταίρων όπως η Κένια και η συνέπεια στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Πρόσφατα συμμετείχα σε μια αποστολή στο Πακιστάν της Υποεπιτροπής μας και διαρκώς είδαμε τα διπλά μέτρα και σταθμά σε ό,τι αφορά τα, τα μη επανδρομένα σκάφη. Δεν μιλάμε για την τεχνολογία μόνο, μιλάμε για ένα πρόγραμμα επιλεγμένων δολοφονιών και θα πρέπει να επιτέλους να ε, το καταδικάσουμε. Να πούμε ότι δεν συμφωνούμε στην Ευρώπη και ότι καταδικάζουμε και τους Αμερικανούς εταίρους μας σε ό,τι αφορά αυτή την πολιτική τους και σε ό,τι αφορά τις βασικές αυτές υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Να σας υπενθυμίσω ότι μέχρι τις 12.30 θα έχουμε διερμηνία. Δέκα λεπτά παραπάνω μας δίνουν οι διερμηνείς. Σας ευχαριστούμε. Τέσσερις συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Να δούμε πόσο χρόνο θα χρειαστούμε. Αλλά σε περίπτωση που δεν πάρετε όλο το λόγο, θα συνεχίσουμε το απόγευμα. Κριστίνα Διπιέτρο, από την Ιταλία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα της δράσης που το Ιταλικό Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. <clears throat> Όταν αντιμετωπίζαμε ένα νομοθέτημα για το 2013, ε, παρουσιάσαμε μια πρόταση η οποία έγινε δεκτή από την Ιταλική κυβέρνηση ως σύστασή μας. Τρία κύρια σημεία νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε σε σχέση με αυτά τα θέματα. Πρώτον, να εξασφαλίσουμε ότι η δραστηριότητα αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης θα πρέπει να είναι σύμμορφη με το Σύνταγμα της χώρας μας και την νομοθεσία μας και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία ε, αντιμετώπισης ασύλου θα πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους και να μην έρχεται σε σύγκρουση με το άρθρο 3 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης να σταματήσει τώρα η διαδικασία της λεγόμενης αναπροώθησης ιδίως και μετά από τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου <clears throat> και ένα τρίτο σημείο είναι να υπάρξει μια ε, προσπάθεια να ξεπεράσουμε τις ε, ρυθμίσεις της οδηγία του Δουβλίνου που λέει ότι το κράτος μέλος πρώτης εισόδου είναι αυτό το οποίο είναι αρμόδιο για να αντιμετωπίσει τις αιτήσει ασύλου. Η μεταρρύθμιση στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο σε σχέση με τη σύμβαση με τους που αφορά τους πρόσφυγες γιατί πολλές φορές ο, ο ετών άσυλο παραμένει σε μια κατάσταση ουσιαστικά ε, ε, μια κατάσταση που δεν μπορεί να βγει από τη χώρα αυτή όπου έχει, έχουν ληφθεί τα, τα δακτυλικά του υποτυπώματα και του απαγορεύεται η δυνατότητα να πάει σε άλλες χώρες όπου θα μπορούσε να τύχει μιας ε, πιο ευνοϊκής μεταχείρισης. Είναι σε μια κατάσταση λοιπόν προσωρινής εξορίας. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό και σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του, των Ηνωμένων Θα πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε το τωρινό σύστημα του Δουβλίνου και θα πρέπει να υπάρξει και μια συνεργασία με όλους τους ε, ε, εμπλεκόμενους και συγκεκριμένα και με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι εδώ παρόντες. Σας ευχαριστώ. ο κύριος Σεφενής και από την Πολωνία. Έχεις Θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ απόλυτα. Είναι απόλυτο το δικαίωμα του, στη ζωή και επομένως όλα αυτά τα πειράματα που έχουν να κάνουν με κλωνοποίηση, με ανθρώπινα έμβρια. Είναι επίσης μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί των ανθρώπων που βρίσκονται σε κόμμα και που μπορούν να περιμένουν κάποια βελτίωση της ζωής τους, ότι αυτοί δεν θα πρέπει να υπόκειται σε ευθανασία. Θα ήθελα να ξέρω αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε θέση να προχωρήσει σε ε, πρωτοβουλίες οι οποίες θα εξασφαλίσουν το δικαίωμα στη ζωή και θα ενισχύσουν τις διατάξεις που το προστατεύουν και ιδίως έναντι των πειραμάτων που γίνονται σε επιστημονικό επίπεδο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σεβερίνσκι. Ο κύριος Νέμετ από την ε, Ουγγαρία. Σας Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Εμείς, στη Δυτική Ευρώπη, στις δημοκρατίες ε, της ε, Δυτικής Ευρώπης, Πώς μπορούμε να παραθέτουμε ε, παραδείγματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν εμείς ε, αγνοούμε το δικαίωμα στον ιδιωτικό βίο και αναφέρομαι στην υπόθεση Snowden και στο γεγονός ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε παρακολούθησαν ε, Ευρωπαίους πολίτες. Συμμετείχε μάλιστα, συμμετείχαν βέβαια και οι Βρετανικές υπηρεσίες σε αυτήν την διαδικασία της παρακολούθησης των Ευρωπαίων πολιτών. Πώς μπορούμε λοιπόν να διακηρύττουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ως Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ε, δεν έχουμε βάλει σε τάξη τα του οίκου μας, πώς ε, ζητούμε από τους Ρώσους εταίρους μας, για παράδειγμα, να σεβαστούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όταν εμείς οι ίδιοι παραγνωρίζουμε σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα εδώ ε, στην Ευρώπη. Ξέρω ότι συζητάτε αυτό το θέμα και ελπίζω να υπάρξει θετική έκβαση στις αυτές. Και τώρα στρέφουμε προς συναδέλφους, προς τα Εθνικά Κοινοβούλια. Παρακαλώ πολύ να τεθεί αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη στις χώρες σας. Ευχαριστώ πολύ αν συμφωνεί ο κύριος Σατούρος από την Ελλάδα, στην επόμενη ε, συνεδρία μας θα ε, σας δώσω το λόγο, για να δώσω το λόγο στον κύριο Τόερμαν να απαντήσει να μας απαντήσετε στους, και στους συναδέλφους ε, από την Ιταλία, αλλά και στο δικαίωμα, στο ιδιωτικό βίο ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια αυτό είναι θέμα που θα μας απασχολήσει και το απόγευμα για τη συνοχή ε, εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο της, των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Τόιερμαν, ευχαριστώ πολύ πράγματι. Είναι γεγονός ότι οι ερωτήματα που μου ετέθησαν ε, θα είναι το αντικείμενο της απογευματινής συζήτηση σε σχέση με τη συνοχή και όπως είπα απαντώντα και στον κύριο Νικολέτη σε σχέση με αυτά που με ρώτησε για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, στην ΚΟΧΟΜ ε, ασχολούμαστε κυρίως ε, με την εξωτερική διάσταση, αλλά κατά το πρώτο ήμιση αυτής της χρονιάς ε, δώσαμε ιδιαίτερες κατευθυντήρες γραμμές για το πώς μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών Επίσης είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την κατάσταση και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως μερικές περιπτώσεις ε, για ε, τις οποίες παρατηρήσαμε εξελίξεις και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο για μας ήταν προϋπόθεση για να έχουμε μια ισχυρότερη θέση έναντι των τρίτων χωρών. Πριν από δύο ε, χρόνια υπήρξαν ε, σημαντικές εξελίξεις, ε, υπήρχαν αποφάσεις από το δικαστήριο και ανάπτυξη νομοθεσίας και πολιτικών σε διάφορα κράτη-μέλη. Είχαμε την ίδια συζήτηση και νωρίτερα αυτή τη χρονιά για τις κατευθυντήρες γραμμές πώς μπορεί να ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ελευθερία των θρησκευτικών πεπιθήσεων. Ήταν μια συζήτηση που ήταν σημαντική και στο εσωτερικό επίπεδο. Υπήρξε σχέδιο δράσης λοιπόν για το πώς μπορεί να ενισχύσει ε, την ε, ε, εφαρμογή δικαιωμάτων στο διαδίκτυο αλλά και εκτός διαδικτύου. Είναι σημαντικό θέμα και η αξιοπιστία των εργασιών μας. Αυτό δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά είναι σημαντική συνιστόσα για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για να σταματήσουν οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμφωνώ όμως απολύτως μαζί σας ότι ο στόχος μας ε, δεν είναι απλές δηλώσεις, αλλά να ε, κάνουμε τη διαφορά. Μερικές φορές χρειάζεται να είμαστε πιο ε, να, να είμαστε πιο επικριτικοί, σε άλλες περιπτώσεις πρέπει να είμαστε πιο διπλωματικοί. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία προσέγγιση. Είναι λίγο διαφορετικές οι προσεγγίσεις μας ανάλογα με το αν πρέπει να ενισχύσουμε τους προασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μερικές χώρες και από πολιτικής απόψης, σε μερικές φορές και χρηματοδοτώντας. Είναι μία από τις προκλήσεις ε, όταν πρέπει να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπό μας ε, στα θέματα αυτά. Μερικές φορές ε, δεν μπορούμε σε μερικούς μήνες να δούμε τα αποτέλεσματα αυτά, πρέπει, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Και είναι δύσκολο κανείς ε, να προσμετρήσει ακριβώς ποιο ήταν το ποσοστό της δικής μας συνεισφοράς. Σε μερικές περιπτώσεις ε, δεν ε, γίνεται τίποτε, αλλά ξαφνικά αλλάζουν τα πράγματα. Πάντως εμείς θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά το σχέδιο δράση και το στρατηγικό πλαίσιο το οποίο ενέκριναν οι υπουργοί, συζήτησαν επίσης το θέμα ε, της εφαρμογής τον Ιούλιο σε ε, συνεδρίασή τους ε, Την πρώτη φορά που ενέκριναν ε, ε, χειροκρότησαν όλοι οι υπουργοί ε, μέσα στην αίθουσα, την πρώτη φορά που ενέκριναν το κείμενο αυτό, κάτι το οποίο δείχνει τη δέσμευση των κρατών μελών στην επίτευξη των στόχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν υπάρξει και πολλές εξελίξεις κατά τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε τώρα πώς θα το εφαρμόσουμε αυτό κατά περίπτωση, γιατί υπάρχουν πολύ διαφορετικοί παράγοντες που το καθορίζουν αυτό και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ε, υπόθηκε επίσης όταν μιλάμε ε, με το θέμα της οικονομικής κρίσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με την οικονομική κρίση. Εμείς ασχολούμαστε κυρίως με την εξωτερική διάσταση, αλλά βεβαίως ε, το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει και το απόγευμα. Υπάρχουν σημαντικές ε, εξελίξεις ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικές πρωτοβουλίες ε, που δεν αποτελούν τμήμα του σχεδίου δράσης γιατί δεν είναι τμήμα του πεδίου εφαρμογή του. Μπορέσαμε όμως, επειδή ετέθη το θέμα αυτό, πώς εξασφαλίζουμε ε, τη σωστή εφαρμογή των κρατών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πώς λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις πολιτικές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αναπτυξιακή, την εμπορική κλπ. Αυτό ήταν σημαντικός στόχος του σχεδίου δράσης και της στρατηγικής. Όλες οι δεσμεύσεις υπάρχουν, πρέπει να ενσωματώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις, τις ε, πολιτικές ένωσης, δεν θα τις αναφέρω επιγραμματικά στην ανάπτυξη, στο εμπόριο, στη δικαιοσύνη και τα εσωτερικά θέματα και πολλούς άλλους τομείς. Πολλή δουλειά γίνεται ήδη. Σε πολλούς από τους τομείς αυτούς ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, κάτι το οποίο είναι σημαντικό όταν ε, καταρτίστηκε το ε, έγγραφο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε και υπήρξε μια πραγματικά ισχυρή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπαιξε και θα συνεχίσει να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία που ήθελα να καλύψω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Τόιρμαν. Και τώρα θα ολοκληρώσουμε την πρωινή μας συνεδρίαση. Ε, περάστε αν θέλετε έξω όπου έχουμε διοργανώσει ένα μεσημεριανό μεσάντουιτς και θα ξαναξεκινήσουμε στις 3.